I think we can start. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Yeah. Ωραία. Καλημέρα. Συνεχίζουμε την ε, συνεδρίασή μας. Αποφάσεις συντονιστών έχουν διανεμηθεί και οι αποφάσεις της τη 9 του μηνό, αν δεν υπάρξουν αντιρρήσει στι 3 το μεσημέρι, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται. Πάμε στι ψηφοφορίε. Να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία πρώτα. Ανοίγει η ψηφοφορία. niemand zu viel. Niemand Pieper ist. So, die Abstimmung hat geklappt. Ωραία. Λειτουργούν όλα άψογα. Όχι, η Γκεζίνα έχει κάποιο προβληματάκι μάλλον. Ωραία, τελείωσε η ψηφοφορία μας. Όλα εντάξει λοιπόν. Λείπει μία κάρτα. Πάμε λοιπόν στην ψηφοφορία για τις διαστάσεις και τα βάρη. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1, τροπολογία 1, corresponding part, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία, γιατί βρισκόμαστε σε δεύτερη ανάγνωση και επιτρέπεται η υποβολή τροπολογιών μόνο από μέλη ή αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Ε, τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Δεν θα τη χρήσει ψηφοφορία. Τροπολογία 8. Όχι, συγγνώμη. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 9 αποσύρθηκε. Πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Συγγνώμη, ξέχασα την κάρτα ψηφοφορία. Θα μου τη φέρει βοηθό. Μπορώ να θεωρηθώ ότι ψηφίζω παρομοίω όπω η συνάδελφό μου η κυρία Αγνοτού. Ναι. Ah. Äh, ja, äh, τη ψηφοφορία, θα την ξανακάνουμε. Έχουμε τρεις, τρία μέλη που δεν έχουν κάρτα ή δεν, ή δεν λειτουργεί η δεν η λειτουργει η καρτα τους. Να σηκώνουν το χέρι τους παρακαλώ. Λοιπόν, ένας ψηφοφορίας τώρα και τα τρία αυτά μέλη να μας πούν τι ψηφίζουν. Υπέρ, κατά, Ωραία, τότε μόνο τα δύο υπέρ. Δύο ψηφί υπέρ. Τέλος της 41 υπέρ. Καμία εποχή. Κύριε Λάιχφριντ, συγχαρητήρια. Ομόφωνα. So, zur nächsten Abstimmung. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία για το EMCA, για την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας στη Θάλασσα. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχή, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται. Ωραία. Οριστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ξεκινά τώρα. Und hat jetzt die Karten, die zwei, die keine Karten haben? οι δύο που δεν έχετε κάρτες, είναι όλα εντάξει υπέρ, Πέρασε τις ψηφοφορίας. 42 ψήφισαν, 36 συν 1, δηλαδή 37 υπέρ, 6 κατά, 0 αποχές και εδώ συγχαρητήρια στον Ντομινίκ Ρικέ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται ε, τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι πρέπει να γίνει έλεγχος. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 5. Ένας ψηφοφορίας. Die Abstimmung ist Πέρας. 33, 34 υπέρ, 7 ε, κατά, εγκρίνεται. Ε, πιο σαφώ σας παρακαλώ να, να σηκώνετε το χέρι σα. Ε, ε, τροπολογία 6. Ε, περ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 7. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Κατά τμήματα υπέρ, για το πρώτο τμήμα κατά, αποχές εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές και εδώ πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Herr Pieper? Okay. ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 17 υπέρ και 26 κατά. τροπολογία 8, όχι, ε, καταπίπτει. Οπότε πάμε στον, ε, στο συμβιβασμό. Συμβαστική πρόταση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχή, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ξεκινά τώρα. Abstimmung μου geschlossen. Τέλος της ψηφοφορίας. 38 υπέρ 5 κατά 0 αποχές. Συγχαρητήρια. Ντομινίκ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ιδεοδρόμων. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική προτάση 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία από την κυρία Γιάλα Σέντερ. Υπάρχουν αντιρρήσει. Τότε ψηφίζουμε μαζί με την προφορική ε, τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οριστική ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία. Ξεκινά τώρα. Πέραση ψηφοφορία. 37 υπέρ, 6 κατά, 0 αποχές. Εγκρίνεται. Για το ΣΕΖΑ ασφάλεια της αεροναυτιλίας. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Με ονομαστική ψηφοφορία, η τελική ψηφοφορία ξεκινά τώρα. Τέλος της ψηφοφορίας. 38 υπέρ 5 κατά εγκρίνεται. Γενικός προϋπολογισμός, απαλλαγή. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. κατά εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 14. 13 και 13 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά. Ξεκινάει τώρα. Τη Τέλος. 37 με έξι εποχές, υπέρ έξι εποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Πυρίνσκι.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 Ja, dann kommen wir zum nächsten. Ε, πάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης. Καλωσορίζω. Την Υφυπουργό Οικονομικών της Λετωνίας, υπεύθυνη για θέματα τουρισμού, την κυρία Ζάγια Λεπίνα. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Σα δίνουμε το λόγο για να μας μιλήσετε για τις προτεραιότητες Λετωνική Προεδρίας στον τομέα του τουρισμού. Καλή σας μέρα. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Κράμερ, αξιότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τα χαράς απευθύνομαι στην Επιτροπή σας και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να αλλάξουμε απόψεις ε, για το θέμα του τουρισμού και να παρουσιάσω τα βασικά θέματα που αφορούν τον τουριστικό τομέα. Θέματα τα οποία θα καλύψουμε στην Προεδρία μας. Στην αρχή του έτους παρουσιάσαμε προτεραιότητες της ε, Λετωνικής Προεδρίας, άλλους τομείς που εμπίπτουν ε, στις αρμοδιότητες Επιτροπής. Αλλά σήμερα θα αναφερθώ στον τομέα του τουρισμού θα αναφερθώ στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευρώπη. Μέχρι 5% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ενώσης αντιπροσωπεύει ο τουρισμός, μαζί με άλλες σχετικές βιομηχανίες, συνεισφέρει σε πάνω από 10% του ΑΕΠ. Η τουριστική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει εργασία σε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ανθρώπους που ασχολούνται σε 1,8 εκατομμύρια εταιρείε. Άρα είναι ιδιαίτερα σημαντικός τομέας για οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η περιοχή στον κόσμο που επισκέπτονται οι περισσότεροι. 40% των διεθνών ταξιδιωτών επισκέπτονται την Ευρώπη. Αλλά για να παραμείνουμε σε ηγετική θέση δεν μπορούμε να αναπαυθούμε στις, να αναπαυθούμε στις δάφνες μας. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν τουριστικού προορισμού και να προσαρμοστούμε στις πρόσφατες τάσεις και προκλήσεις του τουριστικού τομέα. Έχουμε εντοπίσει τρεις βασικές προκλήσεις για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας. Πρώτα μπορούμε να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν προορισμό της Ευρωπαϊκής του τουρισμού, να παράγουμε και άλλα προϊόντα τουριστικά και να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο για, την, για τον τομέα. Μιλώντας για την πρώτη πρόκληση, δηλαδή βελτίωση της θέσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσης σαν τουριστικού προορισμού. Να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από άλλους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Νοτιοανατολική Ασία και η Κίνα. Ο τουρισμός γίνεται όλο και πιο σημαντικός για την οικονομική ανάπτυξη και στο πρόγραμμα της Προεδρίας έχουμε δεσμευτεί να κινηθούμε προς διατήρηση του καθεστώτος Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να εξακολουθεί να είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν τα κράτη-μέλη και να βελτιώσουμε το ευρωπαϊκό όνομα στις ε, αγορές της Ανατολής. Για να ανταγωνιστούμε καλύτερα ε, θα πρέπει ο ευρωπαϊκός τουρισμός να αναπτυχθεί και θα πρέπει να διατίθεται στην αγορά με καλύτερο τρόπο. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβληθεί σαν βιώσιμος τουριστικός προορισμός υψηλής ποιότητας. Η πολιτική ή τουριστική θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των τουριστικών προορισμών και θα πρέπει να υποστηρίξουμε διάφορα διασυνοριακά προγράμματα και διάφορα έργα τουριστικά. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να ε, διεισδύσουμε σε μακρινές τουριστικές αγορές όπως η ΙΠΑ, η Ιαπωνία και η Κίνα είναι να προωθήσουμε την Ευρώπη σαν ενιαίο τουριστικό προορισμό. Να προβάλλεται μια κοινή εικόνα. Έτσι θα προωθείται η Ευρώπη κυρίως και οι μικροί προορισμοί της αγοράς. Θα μειωθεί το κόστος προώθησης και διαφήμισης και θα προβληθεί καλύτερα εικόνα. Είναι σημαντικό να δώσουμε τουριστικές διαδρομές που θα καλύπτουν ε, ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τις κοινέ πολιτιστικές αξίες και την ποικιλομορφία που μας διακρίνει. Όπως τα διάφορα τοπία, η πολιτιστική κληρονομιά, ε, οι κουζίνες των διαφόρων περιοχών Δεύτερη πρόκληση, η ανάπτυξη διαφόρων καινοτόμων τουριστικών προϊόντων. Η Λεπτονική Προεδρία θα εστιαστεί ιδιαίτερα επί της αναπτύξεως της ψηφιακής τεχνολογίας. Η ψηφιακή εποχή έχει δημιουργήσει νέες υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού. Πάνω από 95% των ταξιδιωτών χρησιμοποιούν ψηφιακές πληροφορίες και εργαλεία στα ταξίδια τους. υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι είναι σημαντικοί, όπως η καινοτομία στις υπηρεσίες, χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα. Η ψηφιακή Ευρώπη αποτελεί μία από τι προτεραιότητε της Προεδρίας μας. Και το τέλος Μαρτίου, κατά τη διάρκεια του ατύπου Συμβουλίου Ανταγωνισμού, θα συζητήσουμε την ψηφιακή οικονομία. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνόδου θα συζητήσουμε ζητήματα που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και θα διοργανωθεί και η ψηφιακή συνέλευση τον Ιούνιο. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν την ανάπτυξη και προώθηση του ψηφιακού δυναμικού της Ευρώπης και την ψηφιακή ενία αγορά. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι επιταχύνονται οι εξελίξεις στην πληροφορική και την ψηφιακή τεχνολογία. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση περί αυτού στις επιχειρήσεις που κινούνται στον τομέα. Κυρίως ευαισθητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να τις εκπαιδεύσουμε για τα ωφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας. Δηλαδή ταχύτερες και καλύτερες επικοινωνίες με τους πελάτες, μεγαλύτερες δυνατότητες για συμπράξεις διασυνοριακές και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και ανταλλαγή βέβαια γνώσεων και εμπειριών. Τα τουριστικά προϊόντα θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών. Πρέπει να ακολουθούν τις πρόσφατες τάσεις του τομέα, όπου βλέπουμε περιβαλλοντικά, ε, φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια και πιο προσωπικά διαμορφωμένα. Οι ταξιδιώτες ασχολούνται όλο και πιο πολύ για το οικολογικό τους ίχνος. Γι' αυτό θα πρέπει να παρέχουμε υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον. Μια καλή υποδομή διευκολύνει την ποικιλομορφία των επιχειρήσεων, την πρόσβαση στη φύση, στην πολιτιστική κληρονομιά και άλλους τουριστικούς στόχους και μειώνει την ανθρωπογενή πίεση στο περιβάλλον, μειώνει τον αντίκτυπο επίσης της αλλαγής του κλίματος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν καλύτερα δημιουργώντας δέσμες ε, ομάδες επιχειρήσεων που βελτιώνουν ανταγωνιστικότητα, ε, παραγωγή προϊόντων και καινοτομία. Η Λετωνία θα ακολουθήσει τις πρωτοβουλίες, τελικές πρωτοβουλίας για τη βελτίωση μεταξύ κρατών Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε διάφορους τομείς του τουρισμού. Τέλος, η τελική πρόκληση. Δημιουργία βιώσιμου ρυθμιστικού πλαισίου. Ir maksimāli integrēt arī ar citām ούτω ώστε να αναπτυχθούν βιώσιμες πολιτικές. Αυτές θα πρέπει να συντεριάζουν με άλλες τομεκές πολιτικές όπως το μέτρο των μεταφορών διατηρώντας ε, την ε, πολιτιστική κληρονομιά και τη φύση. Παραδείγματο χάρη βλέπουμε μεγάλη ανάπτυξη στον τομέα των κρουαζιερών στην Ευρώπη και επηρεάζεται η οικονομία από αυτές. Είναι σημαντικό όμως να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, ε, αναπτύσσοντας βιώσιμες και υπεύθυνες υποδομές όσον αφορά τα πλοία. Ε, αναφερόμενοι τώρα στο μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας, συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καθορίσουμε τη νέα τουριστική πολιτική και τις σχετικές ε, προτεραιότητες που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επί ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εργάζονται στον τομέα και βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη του τουρισμού. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις επί Λουξεμβουριανής Προεδρίας στα, στις διάφορες αιτήσεις συναντήσεις για τον τουρισμό το φόρουμ, το ετήσιο τουρισμό. Είναι καλό βήμα αυτό για τις συζητήσεις, για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τώρα αναφερόμενοι στο μέλλον, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ρυθμιστικό πλαίσιο. Πρέπει να είναι ισορροπημένο, να είναι φιλικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αυξάνει τη δυνατότητα διεθνούς ανταγωνισμού. Για την ώρα συνεχίζονται οι προσπαθίες για την οδηγία για τα πακέτα ταξιδίων. Έτσι θα μπορούμε να προστατεύουμε καλύτερα τους ταξιδιώτες στα ταξίδια τους και θα προωθήσουμε και τα συμφέροντα του τουριστικού τομέα. Σχεδιάζουμε να ολοκληρώσουμε τους τριγωνικούς διαλόγους μέχρι την αρχή της τουριστικής περίοδου και κλείνοντας τώρα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία που διευκολύνει ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα θα είναι και φιλική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα μειώνει το ε, διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να ενισχύσουμε και τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού. Γι' αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω το ρόλο της νέας ομάδας κρούσης για τον τουρισμό, της Task Force. Ήδη ανέφερα τη μεγάλη σημασία που έχει ο τουριστικός τομέας για την ανάπτυξη της οικονομίας. Γι' αυτό έχουμε δεσμευτεί να επεξεργαστούμε τις κάτωθοι προτεραιότητες. Διατήρηση και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν τουριστικό προορισμό, Δεύτερο, ανάπτυξη και ανατόμων τουριστικών προϊόντων και δημιουργία βιώσιμου ρυθμιστικού πλαισίου. Αξιότιμη Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και δράτω με τι ευκαιρίε να σας καλέσω να επισκεφτείτε τη Ρήγα στις 15 και στις 16 Ιουνίου ούτω ώστε να συμμετάσχετε στο ετήσιο φόρουμ της Ευρωπα... Στατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βαλτική. Θα υπάρξει μια ξεχωριστή σύνοδο, σύνοδος αφιερωμένη στον τουρισμό, εστιαζόμενη στην πολιτιστική ε, κληρονομιά και στα προστασία των τοπίων στον παράκτιο τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ και Αλυπιένα για την παρουσίασή σας. Ξεκινούμε με τον Βιμ Βαντεκάμπ. Ehm, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Υπουργό. Συγχαρητήρια για αυτήν την ε, περιγραφή της κατάστασης, πληρέστατη και των ε, προτεραιοτήτων μας και του προγράμματός σας. Ελπίζουμε ότι εντός των 4,5 μηνών που μένουν θα μπορέσετε να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Ίσως ήμουν αφηρημένος, αλλά δεν άκουσα καμία αναφορά στην ασφάλεια. Ξέρετε, το περασμένο Σαββατοκύριακο λάβαμε γνώση των διαφόρων στατιστικών στοιχείων και συγκεκριμένα της μείωσης ε, του τουρισμού στο Παρίσι μετά τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις ε, στο Παρίσι. Αναφερθήκατε στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στο οικολογικό αποτύπωμα και θα ήθελα να μας πείτε ορισμένα πράγματα σε σχέση με αυτό το θέμα που ε, ρώτησα. Το είχαμε συζητήσει με τη Λετωνική ο Ισμαήλ Έρτουκ, ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους της ε, ομάδας των σοσιαλιστών για την παρουσία σας. Ισχύει ότι ο τομέας των μεταφορών είναι ευάλωτος διότι ο τουρισμός ε, εξαρτάται και από άλλους, ε, άλλους παράγοντες όπως και η ασφάλεια, όπως είπε και ο συνάδελφός μου, από την κατάσταση, την ε, εικόνα μιας χώρας, ο βαθμός στον οποίο έχει αναπτυχθούν, έχουν αναπτυχθεί οι υποδομές και κατά πόσο προσφέρονται για τον τουρισμό. Όταν έχει κανείς υποδομές φυσικά μπορεί να κατευθυνθούν τουρίστες και σε πολλά μέρη. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό οι υποδομές να προσαρμοστούν και με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη της τουριστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημά μου αφορά περισσότερο την συνεργασία των κρατών μελών. Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη είναι ένας ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός παγκοσμίω. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι πολλοί άνθρωποι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελαν ενδεχομένως να επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά λόγω των ρυθμίσεων που ισχύουν για τις θεωρήσεις δεν μπορούν. Ε, γιατί πολλοί ε, αναγκάζονται να περάσουν μέρες ολόκληρες στις ε, πρεσβείες και τα προξενία για να πάρουν θεωρήσεις για να έρθουν εδώ και έτσι αποφασίζουν να πάνε αλλού. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε πολλά προβλήματα λόγω του γεγονότος ότι αυτό αυτές οι ρυθμίσεις για τις θεωρήσεις αναγκάζουν ανθρώπους να πάνε τελικά στο Μαρόκο, στην ε, την Ισία. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό ε, που χρειαζόμαστε είναι μια χαλάρωση των συγκεκριτικών διατάξεων. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα αποτελέσει κάτι τέτοιο προτεραιότητα της δικής σας προεδρίας να ευαισθητοποιήσετε δηλαδή και τους υπουργούς εσωτερικών προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερο ερώτημα. Είπατε και σωστά ότι χρειαζόμαστε νέα κοινοτόμα συγκεκριμένα είπατε τουριστικά προϊόντα και να τα συνδυάσουμε με την ε, χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα τι εννοείτε. Ε, θεωρείτε δηλαδή ε, ότι θα πρέπει κάθε ένας που έχει ένα smartphone σήμερα να έχει πρόσβαση σε τέτοιες προσφορές. Ποια, ποια, ακριβώς εργαλεία φαντάζεστε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει και πλεονέκτημα έναντι των άλλων περιοχών. Και ε, τέλος, μετεκπαίδευση, κατάρτιση στον τουριστικό τομέα. Ε, πώς φαντάζεστε και σε ποιους τομείς φαντάζεστε ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η μετεκπαίδευση. Ενδεχομένως στον τομέα του, του εφοδιασμού, του logistics θα μπορέσετε να αναλάβετε, έχετε σκοπό να αναλάβετε πρωτοβουλία σε, αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο Ρόμπερτ Τζίλελ. Ευχαριστούμε κύριε Λιωτίνη. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε τις προτεραιότητες της, ε, της Λετωνικής ε, Προεδρίας ε, για τον τουρισμό. Είμαστε υπεύθυνοι για τις μεταφορές και τον τουρισμό. Κυρίως όμως ασχολούμαστε με, τον, με τις μεταφορές γιατί έχει διαφορετικό καθεστώς ε, ως από τον τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να αναφερθώ στην πρώτη προτεραιότητα που αναφέρατε, ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να θεωρείται τουριστικός προορισμός για την Ασία. Πολλοί κόσμος θα μπορούσε να προέρχεται από την Ιαπωνία και άλλες ασιατικές χώρες. Μήπως βλέπετε, ποιοι, μήπως έχετε υπόψη σας ποιοι οργανισμοί θα μπορούσαν ε, να ε, κάνουν διαφορετική προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προορισμό και τι πόρους θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί χωρίς τους πόρους δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, στην Ελβετία υπάρχουν προϊόντα που ε, προωθούνται πάρα πολύ ε, ως ε, συγκεκριμένες οδοί τουριστικές, συγκεκριμένοι προορισμοί. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα σε σχέση με την πρώτη προτεραιότητα που αναφέρατε. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις εξηγήσει. Θέλω να πω ότι καταρχήν συμμερίζομαι τις προτεραιότητές σας και πιστεύω ότι είναι καλά μαντάτα που θέλουμε να προωθήσουμε στην Επιτροπή τον τουρισμό. Ε, ζούμε στιγμές και εποχές ε, όπου είδαμε και στην πρώτερη θητεία ότι ο τουρισμός δεν ήταν προτεραιότητα και δεν μιλούσαμε για την ανάγκη τέτοια σημαντική ανάπτυξη. Σα συγχαρώ λοιπόν για αυτό το νέο βήμα ε, και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ηγετική θέση, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κατάρτιση, να προωθήσουμε την ε, και να αναπτύξουμε την ε, βιωσιμότητα και να προωθήσουμε και το ευρωπαϊκό όνομα και θα πρέπει να προωθήσουμε και ψηφιακά προϊόντα. Και όταν ε, οργανώνουμε την ψηφιακή μας ε, οικονομία Πρέπει να προσπαθήσουμε σε περιοχέ όπω είναι και η περιοχή των Βάσκων να προωθήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία. Έχουμε πολλού τουρίστε οι οποίοι έρχονται στην χώρα των Βάσκων και αυτό είναι πρόσδεκτο. Είναι ένα παράδειγμα που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Μπορούμε να δούμε τι πόροι διατίθενται, να χρησιμοποιήσουμε το βέλτιστο τρόπο τους πόρους. Θα πρέπει να είμαστε σε ηγετική θέση και θα πρέπει να έχουμε και μια δίκαια κατανεμημένη ανάπτυξη τουριστικού τομέα. Πρέπει να έχουμε στόχους και να εξασφαλίσουμε το ότι θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους για να προωθήσουμε τον τουρισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διερωτώμε λοιπόν τι πόρους προτίθεστε να διαθέσετε όσον αφορά την κατάρτιση. και προώθηση του τουρισμού σε λιγότερο ενδειγμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα υπάρξει σημαντική αναπτύξη του αριθμού των τουριστών που θα έρχονται στην Ευρώπη μέχρι το 2030. Δεν θα έπρεπε να δούμε και να εξετάσουμε τη σημασία του εντοπισμού προγραμμάτων με προτεραιότητα και να εξασφαλίσουμε διαλειτουργικότητα στις μεταφορές και να ολοκληρώσουμε τις προτάσεις για τον ενιαίο ουρανό, ούτως ώστε να μην υπάρχουν φραγμοί εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως φόροι, δασμοί, όσον αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια κλπ. Διότι δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι τουρίστες θα έρθουν τα επόμενα 15-20 χρόνια. Ξέρουμε όμως ότι θα αυξηθούν και θα πρέπει να κατανεμηθούν αυτοί οι τουρίστες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και με εκπροσώπους σε άλλους τομείς. Το Συμβούλιο το κάνει αυτό. Εστιάζεται επί της ανάγκης πρόθεσης διαλειτουργικότητας όλων των τομέων. Έχω υπόψη μου προφανώς τις μεταφορές. Θα είναι σημαντικό όμως και για άλλους τομείς. Θέλουμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό και τις μεταφορές. Και θα πρέπει να έχουμε ε, και πιο προχωρημένες μάρκες και ε, καλύτερες προτάσεις ούτως ώστε να προχωρήσουμε όσο πρέπει ολοκληρώνοντας την ψηφιακή αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Μπιλμπάου. Γιατί μιλάμε για τη χρηματοδότηση του τουρισμού και των μεταφορών. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η άποψη της Λετωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αλλάξουμε το κέντρο βάρους της χρηματοδότησης ώστε να λαμβάνεται σοβαρότερα υπόψη και ο τουρισμός και να χρηματοδοτούνται και τέτοιου είδους έργα. Έργα υποδομής δηλαδή που θα επηρεάσουν θετικά τον ε, τουρισμό στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, Καριμαντέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ. Μιλήσατε για αηφόρο τουρισμό μόνο που η κατάσταση σήμερα στον τουρισμό ε, κάθε άλλο παρά φορεία δείχνει. Έχουμε έναν βιομηχανικό τουρισμό ουσιαστικά με κατασπατάληση πάρα, πολλών πόρων ε, ε, και υδάτων ε, και γης. Έχουμε τεράστιο αστικό χώρο που πρέπει να διαχειριστούμε, πάρα πολλές μετακινήσεις. Υπάρχει και ανταγωνισμός σε επίπεδο τιμών που σημαίνει ότι υπάρχει τεράστια αύξηση των οδικών μεταφορών και είναι κάτι το οποίο είναι σε απόλυτη αντίφαση με τους στόχους ε, ε, για τη θέρμανση του πλανήτη. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Σε μερικούς μήνες θα γίνει μια παγκόσμια σύνοδος για την αλλαγή του κλίματος. Ε, τι τι πολιτική θα προτείνετε εσείς και τι στόχους θα προτείνετε κατά τη διάρκεια της ε, προεδρία σας για να ενθαϊνθεί ένας αιφόρος τουρισμός, δηλαδή όλες αυτές οι συνιστώσεις ε, τρόπου μεταφορών που λαμβάνουν υπόψη ε, το θέμα αυτό το ευαίσθητο της θέρμανσης του πλανήτη. Κάτι ακόμη που θα ήθελα να σας ρωτήσω κυρία Υπουργέ, τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσατε γιατί μιλήσατε για την πολιτιστική κληρονομιά, για τη φυσική κληρονομιά, την ιστορική κληρονομιά. Θα ήθελα να μου πείτε για το πρόγραμμα COSME. Τι θα κάνετε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, για τον τρόπο χρηματοδότησής τους και το δεύτερο ερώτημά μου είναι η πρόσβαση όλων στον τουρισμό. Πώς εσείς θα ε, κάνετε προσβάσιμο τον τουρισμό για τους φτωχότερους, για τους ανθρώπους μειωμένη κινητικότητας ή με αναπηρία. Και το τελευταίο ερώτημά μου οι καλές πρακτικές. Εγώ νομίζω ότι ο αηφόρος τουρισμός είναι ένας ε, ήπιος τουρισμός, μία κινητικότητα αηφόρος. Πώς θα το προωθήσετε αυτό, για παράδειγμα με ε, ε ποδηλατοδρόμους και τέτοιου είδους ε, ε, δράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πέτερ να έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Μπερδεύομαι κάπως ακούγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να αναπτύξει τον τουρισμό στην Ευρώπη. Σαν πολίτης αισθάνομαι ότι καθ... οι διαφορές μεταξύ των χωρών, τα χαρακτηριστικά, τα διαφορετικά τοπία ε, οδηγούν στον κόσμο να θέλει να επισκεφτεί διάφορες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πώς μπορεί να βελτιώσει τον τουρισμό υπό οποιαδήποτε μορφή, δεν το καταλαβαίνω. Τι προτίθεστε να κάνετε πάνω σε αυτό. Αν θέλετε να πουλήσετε την Ευρώπη σαν μία μονάδα ενιαία, αν θέλετε να ετοιμάσετε έναν οδηγό στο διαδίκτυο για την Ευρώπη και να παρουσιάζονται οι προσφορές των κρατών μελών, δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω να δω έναν τουρισμό εναρμονισμένο στα κάτι μελη να εναρμονίζεται μέσω κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κάθε χώρα θα πρέπει να μπορεί να διατηρεί τις ιδιαιτερότητες της όσον αφορά τον τουρισμό. Και μπερδεύομαι ακούγοντας τον κύριο Έτσοκ να λέει ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα των ανθρώπων στις θεωρήσεις. Έχουμε τρομοκράτες τώρα, μας βομβαρδίζουν. Έχουμε ε, φρουρούς και έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενόπλους. Εγώ δεν συμφωνώ με τη φιλελευθερωποίηση των θεωρήσεων. Αντίθετα, πρέπει να είναι πιο σκληροί οι κανόνες. Πιο σκληρή έλεγχη στα εξωτερικά σύνορα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε να πηγαίνουν έρχονται ελεύθερα οι διάφοροι. Είδαμε ότι το αποτέλεσμα αυτών ήταν τρομοκρατικές επιθέσεις. Ε, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υφυπουργέ, το 2013 ο αριθμός των τουριστών που επεσκέφθησαν την Πολωνία αυξήθηκε κατά 7%. Σημαντική αύξηση. Πάνω από 15,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Μόνο όμως 90.000, δηλαδή μισό της εκατό ήρθαν στην περιοχή μου. Παρόλο που είναι πολύ ελκυστική περιοχή και πολιτισμικός και άλλος πώς. Υπάρχει και κλειμένος ε, πύργος της πίζας, αλλά υπάρχει και παρόμοιος και στο Τόροιν που είναι η πόλη μου. Και θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη που είναι ελκυστικότατες τουριστικά. Όμως δεν ε, ωφελούμεθα όπως θα έπρεπε από αυτό. Και έχουμε πόρους για προώθηση του τουρισμού. Και έχω αυτή την ερώτηση. Έχετε κάποιες ιδέες για ανάπτυξη του τουρισμού σε περιοχές που είναι ελκυστικές τουριστικά αλλά δεν προσελκύουν τελικά πολλούς τουρίστες. Πρέπει να το προσπαθήσουν αυτό οι ίδιες οι περιοχές ή θα κάνει κάτι η Προεδρία περί αυτού. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μάθω και εγώ πού βρίσκεται αυτός ο κεκλειμένος πύργος της Πολωνίας. Μπορείτε να μας το πείτε στη συνέχεια, κύριε Σισμανουή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία που μας επέτρεψε τη διεξαγωγή της σημερινής συζήτησης χτες Γνώρισα την κυρία φυπουργό και τους συναδέλφους της και διαπίστωσα ότι έχουν πράγματι ε, πιστεί ότι πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες στον τομέα του τουρισμού. Όμως έχω αμφιβολίες όσον αφορά το τι θα καταφέρουμε τελικά. Όχι σχετικά με το τι κάνουμε εμείς στην Επιτροπή μας, αλλά σχετικά με αυτά που γίνονται από πλευράς Προεδρίας. Διότι όταν θα απαντήσει στις ερωτήσεις μας, μέχρι να απαντήσει ερωτήσεις θα περάσει η Προεδρία. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε επί, δύο, ε, ενός ή δύο συγκεκριμένων θεμάτων. Υπάρχουν δύο σημεία που θα ήθελα να τονίσω όσον αφορά τον τουρισμό. Ένα σημείο που το άκουσα και στην παρουσίασή σας και χάρηκα γι' αυτό. Το θέμα του ευρωπαϊκού ονόματος, του brand, της μάρκας συζητείται εκτενώς από τις αρχές των διαφορών χωρών και στο Κοινοβούλιο. Δεν κατανοούν όλοι ότι ο παγκόσμιος τουρισμός άλλαξε. Σαν τομέας άλλαξε. Και όχι μόνο σε ορισμένες περιοχές της ε, Ευρώπης υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους, αλλά υπάρχουν και ήπειροι στον κόσμο που ανταγωνίζονται οι μεν τους δε αυτό το εξάμεινο θα καταφέρετε αυτό το θέμα να είναι συνέχεια στην ημερήσια διάταξη. Όχι μόνο εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά σε κάθε βήμα συζητήσεων. Αφόσον η Ρήγα προεδρεύει, αυτή η ιδέα της μάρκας να είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη. Έτσι θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τους πολιτικούς και για τις επόμενες προεδρίες να αποκτήσει περιεχόμενο αυτή η λέξη μάρκα, brand. Εγώ λέω αυτό το θέμα της μάρκας να το προωθείτε. Διότι αυτό θα το θυμούνται όλοι έτσι και θα το καταναήσουν ακόμα και εκείνοι που δεν το κατανοούν ότι χρειάζεται αυτή η ευρωπαϊκή μάρκα, το brand. Κάτι άλλο τώρα. Αυτό το εξάμεινο, την άποψή μου, είναι ένα εξάμεινο που θα προσελκύσει όλη την προσοχή το πακέτο Juncker και η συζήτηση για την εφαρμογή του προγράμματος. Οι συζητήσεις θα γίνουν περί αυτού και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Εγώ σαν σοσιαλδημοκράτης μπορώ να το δω το πακέτο Juncker με ένα μόνο τρόπο. Δίνει κοινωνική ασφάλεια, δημιουργεί απασχόληση στους Ευρωπαίους πολίτες. Για την ώρα μας ο κύριος Γιούνκερ και οι συνάδελφοί του δεν έχουν κατανοήσει ότι για τον τομέα μας, για τον τουρισμό, η ανάπτυξη του τουρισμού, η λειτουργία του τουρισμού, χρειάζονται υποστήριξη από όλη την Ευρώπη. Διότι συνδέεται το θέμα αυτό με τη δημιουργία της απασχόλησης. Ή, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, με απώλεια θέσεων εργασία. Προτείνω λοιπόν στην Προεδρία να φροντίσει ούτω ώστε όσοι συνεδριάσει του Συμβουλίου, όχι μόνο κατά τη στιγμή που συνεδριάζετε με τους ομολόγους σας, αλλά όταν μιλάτε και σε άλλα βήματα συζητήσεων, όταν συζητάτε για την απασχόληση, για την κατάρτιση, για την εκπαίδευση, κάθε φορά που μιλάτε για το πακέτο Juncker να υπενθυμίζετε τον τουρισμό. Ήδη αυτό θα αποτελεί από μόνο του μια επιτυχία. Αν έχουμε, θέλουμε να έχουμε μια επιρροή ε, όσον στο Συμβούλιο και να μην υπάρχει μόνο η πίεση που ασκείται από τα διάφορα λόμπι εδώ στο Κοινοβούλιο. Το λέω εγώ γιατί προέρχομαι από μια χώρα που είναι κοντά στην περιοχή της κρίσης και επαναλαμβάνω πάντα ότι ο τουρισμός είναι σημαντικότατος. Αυτά και σας ευχαριστώ κύριε Υφυπουργέ. Ευχαριστώ η κυρία Κλάουδια Ταπαντέλα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ε, Φυπουργό που είναι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αναλύσατε τις, ε, προεδρί, τις ε, προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Είναι πολύ σημαντικές και για μας. Είμαι μέλος της Επιτροπής, αλλά είμαι και πρόεδρος της ομάδας προώθησης του τουρισμού. 150 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου, από όλες τι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση συμμετέχουν και από όλες τι πολιτικές ομάδες. Οπότε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα ο τουρισμός για αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Αυτό που με απασχολεί εμένα ως μέλος της ε, Επιτροπής αυτής είναι το εξής. Πρέπει να τονίσουμε τη σημασία των διαφόρων περιφερειών της Ευρώπης. Έχουμε πάρα πολύ όμορφες περιφέρειες και δεν μιλάω μόνο για τις πρωτεύουσες και τις μεγάλες πόλεις. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό στις περιφέρειές μας, το οποίο δεν το αξιοποιούμε γιατί δεν υπάρχει καμία διαλειτουργικότητα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μία λύση. Χρειάζεται βέβαια ε, επενδύσεις και υποδομές. Ένα ακόμη θέμα που θα ήθελα να θέσω είναι κάτι που προέρχεται από την εμπειρία μου στον τομέα του τουρισμού. Έχω παρατηρήσει ότι δεν υπήρξε ο τουρισμός προτεραιότητα για την Ευρώπη Χρειάζεται λοιπόν ένα καλύτερο βήμα για να το συζητήσουμε αυτό και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω ένα ευρωπαϊκό έτος τουρισμού. Και θα ήθελα η Λετωνική Προεδρία, αν μπορεί, να μας υποστηρίξει σε αυτή μας προσπάθεια, γιατί ο τουρισμός δεν είναι απλώς ένας οικονομικός τομέας, είναι και μια κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη γενικότερα. Επίσης, πρέπει να το πρόγραμμα Juncker πρέπει να συμπεριλάβει τον τουρισμό. Δεν το έχουμε δει αυτό ακόμα και θα θέλαμε από κοινού με τη Λετωνική Προεδρία να τονίσουμε περισσότερο αυτό το θέμα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα που θα ήθελα να ε, σας ε, επισημάνω. Τώρα, αυτή τη στιγμή, επικεντρωνόμαστε σε αυτό το νέο είδο τουρισμού, αλλά ο πολιτιστικό τουρισμό πρέπει επίση να είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε πάρα, πολλές, ε, πάρα, πάρα πολλά. Ε, πάρα πολλές τουριστικές ε, περιοχές που θα έπρεπε να προσελκύουν περισσότερους τουρίστες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει καλύτερη προώθηση, κοινή προώθηση, ίσως ε, και ε, μια ευρωπαϊκή, ε, ένα ευρωπαϊκό σήμα, μια ευρωπαϊκή μάρκα. Είναι δύσκολο βέβαια να έχουμε μια ενιαία θεώρηση του τουρισμού, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε μια κοινή προσέγγιση προώθηση του τουρισμού στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ να συνεργαστούμε στενά μαζί σας. Ευχαριστώ. Θα κλείσω τώρα τον κατάλογο ε, ομιλητών. Μόντι, Μάισνερ, Μοντέρο. Δύο λεπτά ο καθένας σας παρακαλώ, γιατί αλλιώς ε, δεν θα προλάβουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο θέματα θέλω να θέσω. Πρώτον, προώθηση της Ευρώπης ως προορισμού. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα και είπατε κι εσείς κύριε Φυπουργέ ότι από αυτό θα επωφεληθούν οι μικρότερες περιοχές και θα ήθελα να μου πείτε πώς ακριβώς φαντάζεστε ότι θα γίνει αυτό. Θα υπάρξει κάποιο ταμείο, από πού θα προέλθει η χρηματοδότηση. Γιατί η ανησυχία μου είναι ότι θα χαθούν οι μικρότερες ε, περιφέρειες και περιοχές στον ανταγωνισμό. Αναφερθήκατε επίσης και στην οδηγία για τα, στην οδηγία για τα ταξιδιωτικά πακέτα και στη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά την απασχόληση στον τομέα του τουρισμού. Εγώ ε, ε κατάγομαι από την Ιρλανδία και εκπροσωπώ τους πολίτες εκεί όπου υπάρχει η, ε, η ανησυχία ότι πολλοί τουρίστες φοβούνται ότι αν ε, φιλοξενούν ε, τουρίστες στο bed and breakfast, στο μικρό τους ε, κατάλημα και συμβεί κάτι στους τουρίστες θα έχουν και εκείνοι ποινικές, νομικές ευθύνες για το τι θα συμβεί στους τουρίστες αυτούς. Η Γκεζίνε Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λεπίνα, ελπίζω να πρόφερα σωστά το όνομά σας. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο παράκτιος τουρισμός. Είμαι και πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής και ασχολούμαστε με την ε, γαλάζια ανάπτυξη, δηλαδή τις δυνατότητες που μας προσφέρει η θάλασσα για το μέλλον. Είπατε και για τις ε, κρουαζιέρες και είπατε ότι είναι ένας ε, κλάδος που αναπτύσσεται, αλλά πράγματι υπάρχει και η πρόβλεψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στο μέλλον θα κάνουν διακοπές στις ακτές. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσει προωθήσουμε τον βιώσιμο τουρισμό στην ε, Γερμανία, στην Βόρεια Θάλασσα. Υπάρχει ε, ταυτόχρονα τουρισμός και ε, ε, οικονομική δραστηριότητα βιομηχανία. Είπατε ε, και για την ε, Λετωνία και για σας είναι σημαντικός ο παράκτιος τουρισμός και θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο βαθμό υπάρχει ανταλλαγή απόψεων με άλλες χώρες που επίσης βρέχονται από θάλασσα, έχουν δηλαδή και παράκτη τουρισμό. Η κυρία Εύανς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υφυπουργέ. Με τα χαράς άκουσα να τονίζετε τη σημασία των μικρομεσαίων και την ανάγκη υποστήριξη που έχουν και πόσο σημαντικές είναι για τον τουριστικό τομέα. Ήθελα να πω κάτι για την πολιτισμική κληρονομιά και το βιώσιμο τουρισμό. Αυτό προφανώς σημαίνει οικονομικά, ε, πολιτισμικά βιώσιμο και από πλευρά τοπίου ε, βιώσιμος τουρισμός. Εγώ εκπροσωπώ την Ουαλία δίγλωση περιοχή. Πολύ συχνά τα ουαλικά ε, που δεν είναι επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν αναγνωρίζονται. Δεν αφορά μόνο την προώθηση και προστασία των γλωσσών το θέμα, αλλά και τις, αφορά και την χρήση των γλωσσών για να συμπεριθούν στη στρατηγική. Η στρατηγική του τουρισμού έτσι θα γίνει αποτελεσματικότερη και κάποιες τοποθεσίες μας θα γίνουν ελκυστικότερες είδατε, εξετάστε κατά κάποιο τρόπο τι γίνεται με τις μειονοτικές γλώσσες, πώς θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν. Να αναφερθώ και σε κοινωνικές πτυχές του τουρισμού. Προσβασιμότητα. Αναφέρθηκε ήδη. Σχετίζεται βέβαια με δημογραφικές αλλαγές και πόσο ελκυστικές είναι τοποθεσίες και πώς μπορούν να τις επισκεφθούν άνθρωποι όλων των ηλικιών και όσον αφορά την οικονομία, αφορά τους εργαζομένους. Ακούσαμε σήμερα το πρωί πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός, ο οποίος ενισχύει την οικονομία και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ξέρουμε ότι πολύ συχνά είναι εποχιακές οι θέσεις εργασίας του τουρισμού. Πώς εξασφαλίζουμε ποιοτικέ θέσεις εργασίας, πώς βελτιώνουμε τις ευκαιρίες να μπορεί να εργαστεί ο κόσμος στον τουρισμό και να μην γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευση. Ευχαριστώ κυρία Λουκασεύσκα Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κυρία Υφυπουργέ, ο τουρισμός είναι σημαντικός για μένα. Ζω σε μια περιοχή, βλέπετε, όπου ε, είναι μικρή τοποθεσία και 80% των κατοίκων εξαρτώνται τον τουρισμό. Κατ' παρελθόν δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν είχαμε ωφεληθεί από τα τοπία μας. Ε, βλέπουμε τώρα ότι αναπτύσσεται ο τουρισμός. Δυστυχώς σε αυτά που μας είπατε δεν άκουσα κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά τον αγροτικό τουρισμό. Δηλαδή μικρές εκμεταλλεύσεις που μπορούν να ε, τροποποιηθούν και να μετατραπούν σε κέντρα αγροτικού τουρισμού. είναι κάτι φιλικό προς το περιβάλλον, ενεργό. Ε, ποια είναι η άποψή σας ήθελα να ξέρω για τον αγροτικό τουρισμό. Και το θέμα προωθήσεως του τουρισμού. Συμφωνώ με εκείνους που λένε ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό χωρίς να τον προωθήσουμε. Μακάρι να είχαμε αυτή την ευρωπαϊκή μάρκα, να υπήρχε, αλλά από αυτά που ξέρω από το Κοινοβούλιο, βλέπω ότι αναφέρουμε μεν τις ιδέες, αλλά αφήνουμε τις περιοχές και την τοπική αυτοδίκηση δεν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Δεν αναφερθήκατε στην ασφάλεια στον τουρισμό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ανέφερε και ο Σβαντερ Κάμπ, διότι χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει κινητικότητα. Δεν αναφερθήκατε και στον τουρισμό ανθρώπων με αναπηρία. Ε, και αυτοί θα έπρεπε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά μας. Δεν είπατε τίποτα για τα ποδήλατα, για την ποδηλασία, για τον οικολογικό, τον περιβαλλοντικά φιλικό τουρισμό. Δεν είπατε τίποτα για τη γενιά των ανθρώπων που είναι πάνω από 50, για τους συνταξιούχους, που γίνονται όλο και πιο κινητικοί και που θέλουν να δουν πράγματα που δεν μπόρεσαν να δουν όταν ήταν νέοι. Το ερώτημα είναι η Προεδρία έχει κάποιες ιδέες για όλα αυτά και πραγματικά ε, ε ελπίζω να τα καταφέρετε όσον αφορά την ευρωπαϊκή μάρκα γιατί είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προκαλείται την περιέργεια κάθε φορά που κάποιος αναφέρεται στην περιφέρειά του και ε, σκέφτομαι κάθε φορά σε ποια να αναφέρεται. Ε, μπορείτε να μας πείτε σε ποια περίπου, σε ποια περιφέρεια αναφέρεστε. Μιλάμε για τα, μιλώ για τα Καρπάθια όρη κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Εκεί υπάρχει το Εθνικό Πάρκο και Στάντ. Λοιπόν, να καλωσορίσω, λέει ο Πρόεδρος, ε, μια ομάδα επισκεπτών της κυρίας Αγιάλα Ζέντερ, της κυρίας Μπιλμπάου, που έχουν προσκαλέσει 15 ανθρώπους από την Ομοσπονδία Οδηγών Λεωφορείων της Ισπανίας. Σας καλωσορίζω και θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε μάλιστα στον τομέα σας και τη συζήτηση για τον τουρισμό. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Η Ζαμπέλ Ντεμόντε έχει το λόγο. Καλημέρα, ευχαριστώ την κυρία Υφυπουργό για την παρουσίαση της. Τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο τουρισμός σίγουρα, όπως ακούσαμε από τις παρεμβάσεις, έχει αυξανόμενη ε, σημασία. Υπάρχει και η διακοινοβουλευτική ομάδα και τα σκφόρς επ' αυτού. Ε, και κινούνται. Αναφερθήκατε εκτενώς σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην ψηφιοποίηση. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτήν. Να επισημάνω κάποια σημεία που κατά την άποψή μου θα πρέπει να εμβαθύνουμε από αυτόν. Την αρχή της μάρκας, του brand και τον ενιαίο ευρωπαϊκό προορισμό. Πιστεύω ότι πέρα από την αρχή των πρωτευουσών θα πρέπει να εισάγουμε και τι πιο άγνωστέ περιοχέ, τη υπαίθρου, τι ορειδές περιοχέ, Διότι έναντι μια εγκατάλειψη συνεχού των περιφερειακών ζώνων σε σχέση με τα αστικά κέντρα, Πιστεύω ότι η έννοια τη ανάπτυξη Ευρωπαϊκή θα πρέπει να ευνοεί επίση και τις οικονομίες αυτέ τι περιοχές που ίσω άλλε εποχε ζούσαν από άλλα πράγματα αλλά σήμερα θα μπορούσαν ήσυχα να παίξουν ένα ρόλο βασικό στον τουρισμό. Θέλουμε να διαφανούν και οι ευρωπαϊκές ταυτότητες, οι πολιτισμικές ταυτότητες, οι παραδόσεις, οι μενοτικές γλώσσες που είναι ένα προϊόν το οποίο θα πρέπει να προσφέρουμε όσον αφορά τις, εκείνους που έρχονται από τρίτες χώρες. Και το θέμα της εποχιακής εργασίας είναι ένα θέμα επί το οποίο θα πρέπει να ε, βασίσουμε τις προσπάθειες για να μπορεί να υπάρχει εργασία όλο τον χρόνο στον τουρισμό. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και τα θέματα των Ευρωπαϊκών Ταμείων και Πόρων. Θέλουμε να βοηθήσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά την ψηφοποίηση. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγάλες ε, δυσκολίες στην πρόσβαση στα ευρωπαϊκά χρήματα και έχουμε ταμεία διατομιακά όσον αφορά ε, έχουν δυσκολία τα μικρομεσαία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά ταμεία μήπως θα μπορούσαμε να προστεύσουμε τη διαδικασία για την πρόσβαση των μικρομεσαίων στην ε, επιχείρηση, ε, συγγνώμη, στην Ευρωπαϊκά Ταμεία και να δούμε ακριβώς και πώς καλύπτουν τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ε, αυτές τις επιχειρήσεις. Ο κ. Γκόλνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο παρατηρήσεις ε, που έγιναν ε, από προηγούμενους ομιλητές ειδικότερα για το θέμα των θεωρήσεων που είναι δύσκολο είναι σαφές ε, ότι μερικές φορές η δύσκολη απόκτηση μιας θεώρησης μπορεί να δημιουργήσει μια τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τουρισμού. Νομίζω ότι ο προκάτοχός μου που, ανα... που επέμεινε στην αναγκαιότητα διατήρησης ενός συστήματος ε, ε, πρόσβασης, ε, άδειας πρόσβασης ε, από ε, κατοίκους κάποιων χωρών για τους λόγους ε, της καταπολέμησης τρομοκρατίας ε, ή για λόγους πολύ λιγότερο σοβαρούς αλλά πολύ πιο συχνούς και που έχουν να κάνουν με το θέμα της ε, παράνομης μετανάστευσης. Μιλάμε πολύ για αυτό το θέμα, για το θέμα αυτών των δυστυχισμένων που προσπαθούν μέσω της Μεσογείου και με κίνδυνο της ζωής τους να μπουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως το θέμα του τουρισμού είναι κάτι διαφορετικό ο, η ουσία της παράνομης μετανάστευσης ε, ε, είναι στο γεγονός ότι πολλοί ε, κόσμος μπαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως τουρίστας, έχει μια περίοδο διαμονή συγκεκριμένη και μετά την εκπνοή της προθεσμίας παραμένει στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και δεν φεύγει ποτέ. Κλάουντια Μοντέρο Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Υφυπουργό. Εγώ είμαι από τη Μαδέρα. Επειδή μας είπατε να λέμε από πού είμαστε, είναι μια άκρος περιφερειακή απομακρυσμένη περιοχή, ε, πολύ τουριστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για τις ε, προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας. Πραγματικά μας περιγράψατε πολύ σωστά την κατάσταση. Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με αυτά που είπαν κάποιοι συνάδελφοι. Ε, τρία σημεία συγκεκριμένα ήταν πιο σημαντικά για μένα. Νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τους νέους επιχειρηματίες που αφοσιώνονται στον τομέα αυτό. Και που θέλουν να καταστούν σε διεθνές επίπεδο πιο ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις τους. Μία ακόμη ερώτηση. Διαπιστώνουμε μία αύξηση της κρουαζιέρας ως ε, είδος τουρισμού και επειδή εγώ προέρχομαι και από την περιοχή που σας είπα, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας. Έχουμε καταγράψει αυτήν την ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας και θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορούμε να τον προσεγγίσουμε αυτό τον τομέα. Κάτι ακόμη είναι η πρόσβαση στον τουρισμό. Πώς έχετε σκοπό να δράσετε και ποια εμπόδια θέλετε να υπερβείτε προκειμένου να υπερασπιστείτε τους ανθρώπους περιορισμένης κινητικότητας, γιατί ο τουρισμός είναι ένας ουσιαστικός τομέας για τις οικονομίες των χωρών μας και ειδικότερα για τις οικονομίες του Νότου, γιατί αυτή η οικονομία του τουρισμού θα μπορούσε να είναι ένας μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Να πω κάτι ακόμη για την Πορτογαλία. Το 2014 τα έσοδα του τουρισμού αυξήθηκαν κατά 12%. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικούς ε, παράγοντες ε, που ε, δείχνουν ακριβώς τη βαρύτητα του τουρισμού. Πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα τουρισμού, όχι μόνο ως εργαστήριο ιδεών, αλλά ως μέσο εξέβρισης των καλύτερων πρακτικών. Και τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι σας εύχομαι κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας και ότι δείξατε την ιδιαίτερη σημασία του τουρισμού ε, και τη σημασία του να γίνει ένας τομέας πάρα πολύ ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ιδού λοιπόν οι ερωτήσεις που σας ετέθησαν. Αναμένουμε τις απαντήσεις σας. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να απαντήσετε εντός 10 Είδατε όμως ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμά στην Επιτροπή αυτή ο Περιμένουμε λοιπόν ε, τις ε, απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Καταρχάς, το θέμα της ασφάλειας, το οποίο έθεσε ο κύριος Φαντερκάμπ και άλλοι ευρωβουλευτές. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει έναν ασφαλή τουρισμό και ο κίνδυνος που σχετίζεται με το έγκλημα θα έπρεπε να μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και εσωτερικά και εξωτερικά η ε, μηχανισμοί επιβολής του νόμου, οι διοκτικές αρχές πρέπει να συνεργαστούν ώστε να καλυφθούν οποιαδήποτε κενά υπάρχουν στο θέμα της ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση χρειάζονται προληπτικά μέτρα και όλοι οι τομείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Όσοι τομείς ε, και όσες πολιτικές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, όπως για παράδειγμα η μεταναστευτική πολιτική, η κοινωνική πολιτική, πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη και να συνεργαστούν. Ω προ τα πρόσφατα γεγονότα στο Παρίσι και τη δράση της Προεδρίας σχετικά, θεωρεί η Προεδρία ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για τον τουρισμό. Δεν είναι ε, κάτι το καινούριο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη κάποια ε, μέσα και στρατηγικές ε, αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Το θέμα είναι πώς μπορούν με πιο ενεργό τρόπο να εφαρμοστούν. Και όπως σας είπα, πρέπει σε δύο επίπεδα να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και σε εσωτερικό επίπεδο αλλά και μεταξύ των εξωτερικών εταίρων της Ένωσης. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το Συμβούλιο Υπουργών στις 12 Φεβρουαρίου ενέκρινε περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ως Προεδρία θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συμπεριλάβουμε το θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν ερωτήματα που έχουν να κάνουν με, την, με τις θεωρήσεις και την ε, ελεύθερη χορήγησή τους. Θα ασχοληθούμε εμείς ως Προεδρία με δύο θέματα καταρχάς, τον κώδικα των θεωρήσεων, όπως επίσης και τις ε, απαιτήσει για τα ταξίδια. Το πρώτο θέμα σκοπό έχει να διευκολύνει τα ταξίδια των τουριστών, όπως επίσης και να απλοποιήσει το νομικό πλαίσιο και παράλληλα να διατηρείται στα εξωτερικά σύνορα η ασφάλεια να γίνεται και μία προσπάθεια διευκόλυνσης ε, της ε, δουλειάς που γίνεται στο πλαίσιο της ε, ζώνης Σέγγεν. Θα προσπαθήσουμε επίσης να σημειώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο και να υπάρξει μία εντολή σε σχέση με το θέμα του κώδικα των θεωρήσεων. Υπάρχει για το θέμα βέβαια της θεώρησης των ταξιδιωτών θέλουμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα με το νομικό κενό που ο κανονισμός Σέγγεν εξακολουθεί να έχει σε σχέση σε σχέση με τις ε, σύντομες, με τις άδειες σύντομης ε, διαμονής, θέλουμε να εκδώσουμε μια νέα, ένα νέο είδος θεώρησης ε, για τους ταξιδιώτες μετά τις 90 μέρες μετά την εκπνοή της προθεσμίας της θεώρησης αυτής δεν μπορεί πια ο κάτοχος της θεώρησης να παραμένει σε αυτό το κράτος μέλος. Η Λετωνική Προεδρία θα προσπαθήσει να σημειώσει πρόοδο όσο το δυνατόν περισσότερο και στο τομέα αυτών και θα εργαστούμε επί της πρότασης αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο, υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες σε σχέση με την ε, ευρωπαϊκή μάρκα, ε, την προώθηση των ε, ευρωπαϊκών περιφερειών, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με αυτό το θέμα. Οι τουριστικές ροές είναι σημαντικές και η κοινή ευρωπαϊκή διάσταση του ευρωπαϊκού τουρισμού είναι σημαντική. Δεν πρέπει να, ανταγωνιζόμαστε, να ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας και να ε, κατασπαταλούμε πάρα πολλούς πόρους για αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν άμεσες προσπάθειες διαφήμιση ολόκληρη της Ευρωπαϊκής Ένωση. και αυτό πρέπει να αντανακλάται και στα προϊόντα που προσφέρουμε οι τουρίστε, πρέπει να γνωρίζουν πώς μπορούν να πάνε από τη μία περιοχή στην άλλη, ε, πώς ε, πρέπει να γνωρίζουν τα καινοτόμα προϊόντα και θα ήθελα να τονίσω τις ε, δράσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει η διαφημιστική εκστρατεία Ευρώπη όποτε είσαι έτοιμος που μέσα σε τρία λεπτά δείχνει τις πιο ε, ωραίες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε όμως να βρούμε και άλλους τρόπους είναι σημαντικό να έχουμε ενιαία φωνή κατά την προσέλκυση τουριστικών ροών στις περιφέρειές μας. Και μετά μπορούμε να επεξεργαστούμε το πώς οι τουριστικές ροές θα, διανέμονται, θα κατανέμονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δείχνουμε ακριβώς την ποικιλοφορία, ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των γλωσσών της, ε, της γαστρονομίας της. ως προς τους ε, οργανισμούς που θα μπορούσαν να εργαστούν για αυτή την προσπάθεια. Η Task Force για τον τουρισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη ενθαρρύνει, προωθεί τη διαφήμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μακρινές αγορές κάνει διάφορες δημοσκοπήσεις και προσπαθεί να καταγράψει τα στοιχεία αυτά. Προσπαθούμε μάλιστα να γίνει στις 22 Απριλίου θα γίνει μια διάσκεψη της Task Force αυτής. Ε, εκεί θα γίνει μια προσπάθεια αύξησης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό ε, και προς το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα υπήρξαν και ερωτήσεις. Υπάρχουν και άλλες ε, πτυχές που θέσατε, όπως για παράδειγμα το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια ενιαία τουριστική πολιτική. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε σχέση με τους πόρους μας και πρέπει να μπορούμε να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι, τα μεμονωμένα μας πλέον εκτήματα. Για παράδειγμα στις βαλτικές ε, χώρες έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι πιο αποτελεσματικό να συνεργαζόμαστε ως βαλτικές χώρες, να εκπροσωπούμεθα από κοινού στα διάφορα, ε, διάφορες εκδηλώσεις για να προσελκύουμε τουρίστες από διάφορες χώρες, να συνεργαζόμαστε με δημοσιογράφους, με ε, διάφορες εταιρείες ε, προώθησης του τουρισμού, του τουρισμού. Όσον αφορά τα θέματα του του, των μεταφορών και ε, το θέμα των ε, κρουαζιέρων που αναφέρατε. Εμείς υποστηρίζουμε τις εργασίες της Ιταλικής Προεδρίας που προσπάθησε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τουριστικών ε, κλάδων. Είναι σημαντικό να φτάσουμε σε μια κατάσταση ενσωμάτωσης του τουριστικού τομέα στην επιμελητία, στις μεταφορές, στο πολιτισμό, όλες αυτές οι διαστάσεις πρέπει να λαμβάνονται από κοινού υπόψη. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί και ε, η δημόσια υποδομή προς όφελος της πολιτιστικής κληρονομιάς γιατί έτσι διατηρείται και οι διατηρούνται και οι τουριστικές ε, ε, ροές και η πολιτιστική κληρονομιά. Να αναφερθώ τώρα στο παράδειγμα που ανέφερε και ο κύριος Κράμερ. Ποδηλατόδρομοι που περνάνε από διάφορες χώρες που περνάει από διάφορες χώρες και που είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Γιατί χρησιμοποιώντας έναν τέτοιο ποδηλητόδρομο, οι τουρίστες μπορούν να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και να βελτιώνουν και την υγεία τους. περνάνε μάλιστα και από παράκτιες περιοχές, ε, πάνω από 500... Ε, Η Λετωνία έχει εκτογραμμή ε, πάνω από 500 χιλιόμετρα και αυτό είναι πάρα πολύ αξιέπαινο. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές οι οποίες είναι εκτός των μεγαλύτερων ε, τουριστικών περιοχών. Υπάρχουν ε, και ζητήματα χρηματοδότησης. Πώς μπορεί κανείς να ενθαρρύνει τον τουρισμό. Υπάρχει το πρόγραμμα COSME, τα διαρθρωτικά ταμεία, με τα οποία μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει τα διάφορα προγράμματα και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχει βέβαια και η εθνική και η περιφερειακή χρηματοδότηση που είναι επίσης απαραίτητες για τη συμπλήρωση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Αναφερθήκατε επίσης ε, στις νομοθετικές πτυχές τη μείωση του διοικητικού άχθους. Συμφωνώ απολύτως και κατά την Προεδρία μας κάνουμε μία αξιολόγηση όλων των νομοθετικών πράξεων και της πρόοδου που σημειώνεται σε αυτές, ώστε να είναι απλούστερες, ώστε να είναι πιο φιλικές προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ώστε να μην επιβαρύνουν το διοικητικό άχθος μιλάμε για την οριζόντια πολιτική και καθόλες όλες τις ομάδες εργασίας προσπαθούμε να αναλύσουμε όλες τις νομικές πράξεις βάσει όλων αυτών των πτυχών που μόλις ανέφερα. Και ναι, η ψηφιακή οικονομία είναι μία από τις προτεραιότητες της ε, Λετωνικής Προεδρίας και είναι σημαντικό για μας όλες οι νέες νομοθετικές πράξεις να αναλύονται και υπό το φως αυτής της ψηφιακής ε, οικονομίας αλλά και της ε, ψηφιακής διαθεσιμότητάς τους. Ε, ελπίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να καλύψω όλες τις πιθανές πτυχές. Σας ευχαριστώ πάντως για την προσοχή σας. Χάρηκα ιδιαίτερα που ήμουν εδώ σήμερα και που μοιράστηκα μαζί σας ε, το πρόγραμμα της Προεδρίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και εμεί χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το γεγονό ότι ήρθατε εδώ, το γεγονό ότι μα μιλήσατε. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ο τουρισμό έχει πολλέ διαστάσει και ελπίζουμε να κάνουμε μεγάλα βήματα προ τα εμπρό. Ευχόμαστε σε εσά και στη Λετωνική Προεδρία φυσικά κάθε επιτυχία, γιατί είναι άλλωστε και η πρώτη φορά που η Λετωνία ε, προεδρεύει του Συμβουλίου ελπίζουμε λοιπόν σε μια καλή συνεργασία, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε και πάλι. So, dann zum... Ωραία. Πάμε στην επόμενη, στο επόμενο θέμα της ημέρησης διάταξης, το 17. Καλωσορίζουμε τον ε, κύριο Μπρόινιξ, εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος So, ich glaube, dann können wir anfangen. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλωσορίζω λοιπόν θερμά τον κύριο Μπροενίξ για τις επιπτώσεις τις περιβαλλοντικές πιέσεις προκαλούνται από τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Είναι θέμα που μας απασχολεί. Έχουμε διάφορες απόψεις και για τις συνδέσεις μεταξύ Βερολίνου Μπρέσλαου και άλλες διαδρομές. Θα θέλαμε λοιπόν σε πρώτη φάση να μας πείτε για τις ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων. Ευχαριστώ πολύ που μείνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω το έργο της υπηρεσίας μας όσον μεταφορές και το περιβάλλον. Θα ξεκινήσω... Πού να δείξω, τι να πατήσω το... Yes. Um, e λοιπόν, ο οργανισμός μας έχει μακρά παράδοση όσον αφορά τις μεταφορές και το περιβάλλον. Από το 2000 παράγουμε τήσια έκθεση περί μεταφορών και περιβάλλοντος. Φέτος είναι η 15η επέτειος της εκθέσεως. Στην έκθεση για το 2014 που θα παρουσιάσω σήμερα συλλέγουμε πληροφορίες. Αξιολογούμε το μεταφορικό τομέα όσο σχετίζεται με στόχους και πρόοδο που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά. Προφανώς οι περισσότεροι στόχοι έχουν διατυπωθεί στα πλαίσια της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές. Βλέποντας μακροπρόθεσμους στόχους για το μεταφορικό τομέα και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, βλέπουμε ότι μέχρι το 2050 στόχος είναι να μειωθούν αυτά τα αέρια κατά 60% εν συγκρίση με το 1990. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα, όσον αφορά το ποσοστό αερίων του θερμοκηπίου, ο μεταφορικός τομέας αντιπροσωπεύει περίπου 25%, ακριβέστερα 24,3% όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Εν συγκρίση με το μεταφορικό τομέα, αν συγκρίνουμε άλλους τομείς με το μεταφορικό, ή βλέπουμε ότι είναι ο μόνος μεγάλος οικονομικός τομέας από το 90 όπου οι κομμές αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν. Είμαστε τώρα περίπου 20% πάνω από το στόχο του 90. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη, η συνολική οικονομία έχει μειώσει κατά 20% την εκπομπή αυτών των αερίων. Από το 2007-2008 είδαμε αλλαγή της τάσης και υπάρχουν τρει βασικοί λόγοι γι' αυτό. Σημαντικοί λόγοι που ενδιαφέρουν την Επιτροπή σα. Πρώτον, μετά την οικονομική κρίση βλέπουμε μείωση στη ζήτηση μεταφορικών μέσων, τουλάχιστον σε κάποια μέρη της Ευρώπης. Δεύτερο, αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικών, όπως μέτρα για την αποδοτική χρήση των καυσίμων που ισχύουν έκτοτε και έχουν τα αποτελέσματα που θα δείξω αργότερα. Τρίτον, αρχίζουμε να παρατηρούμε αλλαγή συνθήκων καταναλωτών, συνηθιών καταναλωτών. Κυρίως οι νέοι σταστικά περιβάλλοντα αλλάζουν συνήθειες. Πάμε τώρα στους άλλους στόχους στην Ευρώπη, στο μεταφορικό τομέα, που σχετίζονται με το 60% των εκπομπών. Βλέπουμε ότι μέχρι το 2050, το 2050 στα διεθνή ε, φορτηγά πλοία θέλουμε μείωση το 40% σε σχέση με το 2005 και πιο βραχυπρόθεσμος στόχου θέλουμε 10% ανανεωσίμων πηγών ενεργείας που θα καταναλώνονται μέχρι το 2020 από το μεταφορικό τομέα. Έχουμε τα αυτοκίνητα και τους κανόνες και για τα νέα ε, φορτηγάκια θέλουμε 95 και 147 γραμμάρια ανά ε, χιλιόμετρο στις εκπομπές. Τώρα πηγαίνοντας στο μεταφορικό τομέα, ε, βλέπουμε ότι είναι πολυσχηδής τομέας μπορεί να μοιραστεί επικοιλωτρόπως. Μία διατομή κάνει διάκριση μεταξύ μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών. Στην Ευρώπη περίπου 42% του μεταφορικού τομέα αφορά τα εμπορεύματα και περίπου 60% αφορά τη μεταφορά επιβατών. Αν δείτε τους ε, αριθμούς, είναι αρκετά αξιοσημείωτο το ότι 25% περίπου όλων των μεταφορών ε, παράγεται εντός των αστικών περιοχών και ξέρουμε από διάφορες μελέτες ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αυτό το 25% να μετακινείται ε, προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με τα μέτρα. Να αυξάνεται να μειώνεται ανάλογα με τα μέτρα των πόλεων. Ένα σημαντικό νομοθέτημα βλέποντας την αποδοτική χρήση της ενέργειας στο μεταφορικό τομέα. Και μάλλον ήταν και επιτυχία. Είναι οι μέσες εκπομπές για τα νέα όπου δύο χρόνια πριν από το στόχο μας η αυτοκινητοπιμηχανία της Ευρώπης κατάφερε να πετύχει το στόχο για το 2015. Είμαστε στα 127 γραμμάρια. Ο στόχος ήταν 130 στα, μέχρι το 2015. Και αν συνεχιστεί αυτή η τάση για το στόχο του 2020 μπορούμε να πετύχουμε το στόχο των 95 γραμμαρίων διοξιδιτού άνθρακος ανά χιλιόμετρο. Ποια ήταν μια από τις ανησυχίες που αναφέρουμε στην έκθεση. Είναι από εργαστηριακές συνθήκες πώς αυτά μεταφράζονται σε πραγματικές επιδόσεις στον δρόμο. Για μικρότερα αυτοκίνητα μπορούμε να έχουμε 20 με 25% διαφορά και για μεγαλύτερα οχήματα η διαφορά μπορεί να φτάσει και 30% ή το 1 τρίτο της κατανάλωσης του καυσίμου. Θέλουμε να δείξουμε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κερδών λόγω αποδοτικότητας και γενικής μείωσης των πόρων. Η Ευρώπη ήταν πάρα πολύ επιτυχής όσον αφορά τη μείωση, την αύξηση της αποδοτικότητας των καυσίμων στις μηχανές εσωτερικής καύσεως αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερα αυτοκίνητα και φωτικά στον δρόμο, περισσότερα χιλιόμετρα που οδηγούνται, έχουμε και την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη που κινείται παράλληλα και γενικά λόγω όλων αυτών αυξήθηκε η χρήση των πόρων στο μεταφορικό τομέα. Και εδώ πικονίζεται πολύ σωστά η ε, προσέγγιση με βάση την αποδοτικότητα σε σύγκριση την προσέγγιση με αποδέσμευση των συναφών στοιχείων όπως αφαίρουμε στην έκθεση άλλη επιτυχία λόγω πολιτικών. Αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές στις μεταφορές στην Ευρώπη οδήγησαν και στα άλλα ωφέλη όσον αφορά ρηπαντές, εκπομπή ρηπαντών. Βλέπουμε γενική μείωση της ρήπανσης από δικές μεταφορές. Όσον αφορά τα σωματίδια, 2,5 σε οξύδια του αζότου ε, και πτυτικά ε, πτυτικές ουσίες και οξύδια του θείου. Η μόλι εξαίρεση στη μείωση μέχρι τώρα ήταν ε, ο τομέας των αερομεταφορών λόγω ταχύτητα της αύξησης της ζήτησης. Εν γέννη όμως οι πιέσεις επί του περιβάλλοντος λόγω των μεταφορών όσον αφορά τους διάφορους ρηπαντές έχουν μειώσει. Και αυτό είναι κάτι που απορρέει από την νομοθεσία. Όταν θεσπίζει κανείς νομοθεσία στον μεταφορικό τομέα είναι σημαντικό να κάνει διάκριση μεταξύ μεταφοράς επιβατών και φορτίων. Διότι ο αντίκτυπος είναι διαφορετικός όσον αφορά διάφορους περιβαλλοντικούς ρηπαντές. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά να σας πω ότι όσον αφορά οξύδια του θείου μεταφορά των εμπορευμάτων είναι υπεύθυνη για πάνω από 95% του τυχτυπού. Αν δούμε εκπομπές του άνθρακος, είναι τα πιβατικά οχήματα. Άρα χρειάζονται διαφορετικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις για να πετύχει κανείς αποτελέσματα. Παρά τις μειώσεις. Όσον αφορά τα σωματίδια και άλλους ρηπαντές, ξέρουμε ότι 3 στους 10 Ευρωπαίους που ζουν σε αστικά περιβάλλοντα ζουν σε μέρη όπου έχουμε υπέρβαση των καθημερινών ημερησίων ορίων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και αν πάμε και στην Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στα όρια αυτά, περίπου 9 από τους 10 Ευρωπαίους σε αστικά περιβάλλοντα ζουν σε αυτό πάνω από τα όρια. Παρόλο που έχει πρόοδος, αν δούμε θέματα περιβαλλοντικής υγείας, υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτιώσεων. Τώρα, ένα από τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον είναι τα οχήματα χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα. Βίο, δίζελ, ε, υγρό, αέριο, ε, υβριδικά αυτοκίνητα που είναι μόνο 0,5% των νέων καταχωρήσεων οχημάτων στην Ευρώπη. Όμως αν δούμε τα μέλη της ΕΟΧ που συμμετέχουν και χώρες όπως η Νορβηγία είναι πάνω από 10% για την ώρα. Οπότε είναι 20 ο μέσος όρος της ε, ευρωπαϊκός. Είναι θέμα πολιτικής που μπορεί να επηρεάσει τα μάλα ε, αυτούς τους τομείς τους μεταφορικούς όσους έχουν σήμερα. Η μεγάλη πτώση όσον αφορά τα ε, αυτοκίνητα με υγροποιημένο αέριο οφείλεται σε αλλαγή πολιτικών. Κάποιες από τις μεγάλες χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία αποφάσισαν περίπου το 2008-2009 να μετακινήσουν τους οικονομικούς μηχανισμούς στηρίζοντας το υγροποιημένο αέριο στα καύσιμα και η πολιτική παίζει ρόλο όσον αφορά τις πολιτικές, όσον αφορά το μεταφερικό τομέα. Αν δούμε στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, που είναι περίπου 75% της μεταφοράς φορτίων, πρωταρχικά εξετάζουμε θέματα διεθνών αερομεταφορών και θαλασσίων μεταφορών, όπου έχουμε εδώ 20% όλων των εκπομπών οξυδίων του άνθρακο, περίπου 70% οξυδίων του θείου, και 11% των σωματιδίων 2,5% και αν δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις διεθνείς αερομεταφορές, το 2050 όλα αυτά μπορεί να τριπλασιαστούν. Αν θέλουμε να συμφιλειωθεί αυτό με τη μείωση του 60% στα αέρια του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, υπάρχει ένα σαφές μήνυμα που απορρέει. Πρέπει να αλλάξουμε τη τάση. Τώρα, βλέποντας ποιοι είναι οι παρόντες στόχοι και αν τους βάλουμε σε γραφική παράσταση 2015-2017, νέα οχήματα και τις σχετικές οδηγίες. Έχουν πετύχει τους, ε, κινούμεθα προς τους στόχους. Αν δούμε το 2020-2030 στόχους για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις μεταφορές, αέρια θερμοκηπίου, τα νέα οχήματα, ε, Πομπές διοξιδί του, ανθρώ, άνθρακος, επιμελητία κλπ. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Το ερώτημα όμως είναι τι γίνεται μακροπρόθεσμα. 2050 και μείωση αερίου του θερμοκηπίου κατά 60% στον τομέα κινητικότητα και μεταφορών. Για να πετύχουμε τους στόχους πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από βελτιώσει στην αποδοτικότητα. Αν δείτε τι γίνεται, ε, πόσα καύσιμα έχετε, τα καταφέραμε πολύ καλά να πηγαίνουμε πιο περισσότερα χιλιόμετρα με τέτοια κάψιμα. Βλέποντας τις νέες τεχνολογίες, αν εστιαστούμε επί ηλεκτρικών αυτοκινήτων, βλέπετε εδώ το Τέσλα. Το μεγάλο όνειρο του ηλεκτρικού οδηγού. Είναι η φαντασίωση του κάθε οδηγού που θέλει να οδηγήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι τεχνολογική επανάσταση. Αν οδηγούμε όλοι το ίδιο Τέσλα με τον ίδιο τρόπο, ταυτόχρονα με την ίδια μεταφορά η Ρίντε Λαλουά που όλοι ξέρετε, πάλι 16 ώρες την ημέρα θα είχε τέτοια μορφή. Και θα δημιουργούσαμε άλλα θέματα πόρων, διότι οι μπαταρίες απαιτούν πόρους που δεν έχουμε στην Ευρώπη. Αυτό σας δείχνει ότι για να πετύχουμε μακροπρόθεσμους στόχους χρειαζόμαστε σωστή μετάβαση. Πρέπει να επανεξετάσουμε τα συστήματα Ποιες ανάγκες υπάρχουν. Ποιος είναι ο ρόλος του αστικού σχεδιασμού. Ποιες είναι οι κοινωνικές λειτουργίες σε μια πόλη. Τι γίνεται με τη χωροταξία. Τι αυτοκίνητο θέλει κανείς στην πόλη ή στο αστικό περιβάλλον. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Πώς το χρησιμοποιεί. Ποιες ώρες. Ποια είναι η στο αστικο περιβαλλον ποιος ειναι ο ιδιοκτητης πως το χρησιμοποιει ποιες ωρες ποια ειναι η Και στο τέλος θέλει ένα αυτοκίνητο κανείς που έχει μηδενικές εκπομπές. Άρα σημαντικότατη η τεχνολογία. Αν θέλετε όμως να μην εκπέμπεται άνθρακα στη κινητικότητα και στις μεταφορές, χρειάζεται κάτι πιο σημαντικό. Απαιτεί το ληστική προσέγγιση. Κλείνοντας, θα δείξω δύο διαφάνειες. Η μία αναφέρεται σε μία έκθεση που ετοιμάσαμε. Όσον αφορά την προσαρμογή των μεταφορών στην αλλαγή του κλίματος στην Ευρώπη, δεν θα μακρηγορήσω. Οι μεταφορές και η κινητικότητα πρέπει να πω είναι πολύ σημαντικά θέματα για την Ευρώπη και για την ευημερία των ανθρώπων και για την οικονομία. Περιπλοκότατο θέμα. Εξαρτάται από τεράστιες υποδόμες, τεράστιο κεφάλαιο, ύψιστη τεχνολογία. Αλλά θεωρούμε ότι είναι αρκετά εύθραυστος ο τομέας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος. Αν θέλουμε μακροπρόθεσμο όραμα όσον αφορά τις μεταφορές και την κινητικότητα, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε σε κάποια μέρη της Ευρώπης όπου θα έχει μεγάλο αντίκτυπο ελεγγύη του κλίματος όσο αφορά το μεταφορικό σύστημα αυτά τα στοιχεία να τα λάβουμε υπόψη. Τέλος. Να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα σαν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος θα παρουσιάσουμε την έκθεση που ετοιμάζουμε κάθε πενταετία. Ποια είναι η κατάσταση και το μέλλον για το περιβάλλον. Διαθέτουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε θα το κάνουμε αυτό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μπένεντικ Ζαβόρ, Ζωζέ Ιχνάφιο Φαρία και ο Γιώ Λάινεν διοργανώνουν, συνδιοργανώνουν τη συνεδρίαση αυτή την επόμενη εβδομάδα. Ετοιμάζουμε διάφορες εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες γιατί με αυτό είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε για να σας παρουσιάσουμε ποια είναι η σημερινή και μελλοντή κατάσταση όσον αφορά το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Είστε άκρος ευπρόσδεκτοι να παραστείτε σε αδίποτε τέτοια εκδήλωση. Κύριε Πρόεδρε, εδώ σταματώ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να παρουσιάσω το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Μπρόενιξ για την έκθεση. Υπάρχει και μια μπροσούρα που έχει διαναμηθεί. Μπορείτε να δείτε και εκεί λεπτομερώς τα στοιχεία και θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονό ότι τονίσατε πόσο σημαντικός είναι ο κλάδος των μεταφορών. Εγώ πάντοτε λέω ότι χωρίς αλλαγή της κινητικότητας δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και είπαμε ότι αν, είπατε κι εσείς ότι αν απλώς αντικαταστήσουμε τα αυτοκίνητα με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πάλι δεν θα καταλήξουμε στο στόχο μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι βεβαίως και οι τεχνολογικές ε, εξελίξεις, αλλά και η συμπεριφορά και νομίζω ότι μπορούμε να προστατεύσουμε και την κινητικότητα και το κλίμα. Μπορούν να συνδυαστούν. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση. Ίσως ο κύριος Βινφαμ Ντεκάμπ. Πρώτος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ αναλυτική παρουσίαση των πορισμάτων σας. Γνώριζα ότι ε, έχουν, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά στον τομέα των μεταφορών, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σε αντίθεση όμως με τον ε, Πρόεδρο βλέπω περισσότερες ευκαιρίες παρά απειλές. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε. Έχω μοτοποδήλατο εγώ, οπότε ενδεχομένως ε, δεν έχω δικαίωμα να μιλώ γιατί ε, είναι πολύ ε, ρηπογόνα τα μοτοποδήλατα, ιδιαίτερα αν, όταν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του τουρισμού. Αλλά στην αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε στην αστική κινητικότητα. Νομίζω ότι η αστική κινητικότητα πρέπει να υποβληθεί σε μια ολοκληρωμένη αλλαγή. Υπάρχει μια σειρά ε, προτινόμενων ε, αλλαγών που έχει προτείνει η ε, Παγκόσμια Ομοσπονδία Μεταφορών. Αν δείτε πόσοι άνθρωποι πλέον ζουν σήμερα σε πόλεις με μεγάλα προβλήματα ρήπανσης, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ε, πάρα πολλές αλλαγές. Δεν ξέρω ποιος, είναι, ποιος τελικά είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται. Αναφερθήκατε στα αυτοκίνητα, δεν είπατε όμως για τα τρένα, ε, φορτηγά... εσωτερικές πλωτές οδοί, αεροπορία, αερομεταφορές. Υπάρχουν πολλοί κλάδοι, αλλά γνωρίζουμε ότι οι κινητήρες που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες πλωτές οδού χρησιμοποιούνται για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποιος τελικά ευθύνεται για τη ρήπανση. Να κάνω και, μια, ε, και ένα σχόλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Παρισιού απαγόρευσε όλα τα οχήματα άνω των 20 ετών από την κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Ε, εκτός από συλλέκτες βεβαίως, ε, οι συλλέκτες μάλλον ε, αντικών οχημάτων ε, ε, είναι ανήσυχοι. Μπορείτε να μας πείτε, αλλά ισχύει και για τους... Ε, ε, μπορείτε να μας πείτε τι, την άποψή σας Χαίρομαι που είστε εδώ, γιατί συνήθως όλα τα ζητήματα περνούν μέσα από την Επιτροπή ΕΜΒΙ αλλά θεωρώ και ότι και, εγώ, και, ότι και εμείς ε, ε, είμαστε πολύ ε, σημαντικοί σε αυτό το θέμα. Ο Ισμαήλ Έρτουγκ. Ευχαριστώ κύριε Μπρόνιξ και εκ μέρους των σοσιαλιστών. Πολύ εντυπωσιακά τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Δεν είναι νέα βέβαια, αλλά είναι χρήσιμο να υπενθυμίζονται. Κύριε Μπρόνιξ, είπατε σωστά. Να σας πω ότι έχω οδηγήσει ένα τέτοιο ε, αυτοκίνητο Τέσλα. Αναφερθήκατε σε πολλά θέματα. Θέλω να τοποθετηθώ και εγώ. Και να κλείσω και με μια απέτηση. Μιλήσατε για μια μακροπρόθεσμη προοπτική που χρειαζόμαστε στον τομέα της κινητικότητας. Συμφωνώ απόλυτα είναι ένα θέμα που μας λείπει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το έχουμε επεξεργαστεί ολοκληρωμένα. Και νομίζω ότι ε, πρέπει να απευθυνθούμε και στα κράτη-μέλη, γιατί πολλές φορές τα κράτη-μέλη είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είπατε για το 0,5% των νέων καταχωρήσεων αυτών των ε, εναλλακτικών οχημάτων. Ήμουν σκιώδης εισηγητής για, στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία για το ε, θέμα αυτό και μπορώ να σας πω από τους τριμερούς διαλόγους πόσο δύσκολο ήταν ε, η, πρόταση, η αρχική πρόταση της που θεωρώ ότι ήταν και πολύ καλή πόσο δύσκολο τελικά ήταν να καταλήξουμε σε συμφωνία με τα κράτη-μέλη. Όλες οι δεσμευτικές, ε, όλες οι δεσμεύσεις αντιμετωπίζονται ως... Ε, μεγάλο πρόβλημα ε, για, από τα κράτη-μέλη. Τελικά καταλήξαμε στο, στην θέσπιση ορισμένων μεταβοτικών περιόδων για να καταλήξουν και να επιτύχουν και τα κράτη-μέλη σε κάποιους στόχους. Τα λέω αυτά γιατί ε, αναφερθήκατε και στις εκπομπές οξυδίων του θείου και του αζότου στις αερομεταφορές. Αυτό που μας λείπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, είναι πώς να το πω, δικό χάρτη, master plan. Αυτό που μας λείπει είναι μια συνολική προσέγγιση της κινητικότητας στην Ευρώπη, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλους τους τρόπους μεταφορών και θα λαμβάνει υπόψη το κόστος, τις εκπομπές όλα αυτά τα θέματα. Ανεξάρτητα με, το, με ποιους ενδιαφερόμενους μιλάμε, από παντού τίθεται το ερώτημα ποιος ε, τελικά υφίσταται τα μειονεκτήματα, είτε μιλάμε για τη συνεισφορά για την κυροζήνη, είτε για... Αυτό που μας χρειάζεται είναι μια εποπτεία, να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση αυτήν την συνολική εικόνα να μπορέσουμε να θεσπίσουμε την κατάλληλη νομοθεσία. Αυτό συνέβη εν μέρη και κατά την ε, τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σαφή απάντηση ποιοι τρόποι θα πρέπει να ενισχυθούν ως, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα απαντήσαμε σε αυτό το ερώτημα με τους ιεροδρόμους και με τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Και τα τελευταία χρόνια εκφράστηκαν διάφορες ε, ανησυχίες και προβληματισμοί γιατί δεν, ε, δεν συμφωνούσαν πάντοτε οι προτάσεις των γενικών διευθύνσεων με αυτήν την ε, κατεύθυνση. Άρα, χρειαζόμαστε φυσικά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα Χρειαζόμαστε ενίσχυση της κατανάλωσης, χρειαζόμαστε τις νέες ε, τεχνολογίες, είτε μιλούμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είτε για νέες μορφές αερίου, επενδύσεις ή τρόπους αποφυγής, ε, κατανάλωση καυσίμων, car sharing, κοινή χρήση αυτοκινήτων. Και νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ενισχυθεί και ο αστικός σχεδιασμός. Γιατί τελικά δεν έχει νόημα να... Ε, ε, δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση αν δεν υπάρξει και μετάφραση, μετουσίωση αυτής της συνολικής εικόνας στα, στις πόλεις, στο τοπικό επίπεδο. Είπατε επίσης για, τον, ε, για τις ε, μεταφορές, τις αστικές μεταφορές Τους στόχους μας δεν θα μπορέσουμε να τους επιτύχουμε αν δεν μειώσουμε τις ε, εκπομπές εντός των πόλεων. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιο είδους ε, χρέος, κάποιο είδος χρέωσης για τις αστικές μεταφορές. Σε κάθε περίπτωση η αριθμή που μας παρουσιάσατε είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και είναι σαφές ότι πρέπει να ξεκινήσει μια νέα εποχή. Η είναι Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Κάποιε συμπληρωματικέ παρατηρήσει θέλω να κάνω και εγώ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ακούστηκαν ήδη. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό να ανταποκριθούμε στις ε, αυξανόμενες ανάγκες των μεταφορών. Ξέρουμε ότι οι μεταφορές θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Εμείς θα πρέπει να δούμε πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές και για παράδειγμα είναι σημαντικό να δούμε ε, τι βελτιώσεις μπορεί να γίνουν σε κάθε ε, επιμέρους τρόπο ε, μεταφορών. Θα υπάρξει και αύξηση των οδικών μεταφορών, γιατί δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν όλες οι μεταφορές στους δρόμους και στις πλωτές οδούς. Άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε από οικολογικής άποψη και τι οδικές μεταφορές. Το, αποδείξαμε αυτό και στο θέμα των φορτηγών. Επίσης, ευφυεί συστήματα μεταφορών. Το είπατε κι εσείς. Δεν έχουμε ε, μποτιλιαρίσματα μόνο στις πόλει, πόλεις, αλλά και στις, αυτοκινητόδρομου. αυτοκινητόδρομους. Υπάρχει, για παράδειγμα, στην περιφέρειά μου, ε, ο αυτοκινητόδρομος Α2 αν ε, με έναν έξυπνο τρόπο διαχείρισης μπορούν να αποφευθούν πάρα πολλά μποτιλιαρίσματα. Όπως είπε και ο κύριος Έρτουγκ, ήμουν και εγώ σκιώδης στο πακέτο για την καθαρή ενέργεια. Πρέπει να δούμε ότι ε, οι στόχοι που τέθηκαν ήταν ε, μάλλον όχι ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Η ηλεκτρονική κινητικότητα. Πολύ χαμηλό ποσοστό ακόμη, πρέπει να αναπτυχθεί. Σχετίζεται και με τις υποδομές για την καθαρή ενέργεια, αλλά επίσης σημαντικό είναι από πού προέρχεται αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα. Είδα ένα θετικό παράδειγμα ε, πρόσφατα και μου αρέσει να αναφέρουμε σε θετικά παραδείγματα. Στο Ανόβερο, στο κταίο, ε, προσφέρεται ε, δωρεάν ε, ηλεκτρική ε, ενέργεια για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η οποία μάλιστα η ηλεκτρική ενέργεια έχει παραχθεί αποκλειστικά από ηλιακά πάνελ. Είναι ένα παράδειγμα, για παράδειγμα, και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επαναληφθεί και να το μιμηθούν και άλλες πόλεις, να εγκαταστήσουν δηλαδή πόλεις ε, φωτοβολταϊκά συστήματα και από αυτά να τροφοδοτούνται μετά ε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Βιωσιμότητα, φυσικά το είπαμε, ε, υπάρχουν και στις Βρυξέλλες για παράδειγμα και στο Μεξικό όμως που βρέθηκα πρόσφατα πολλά ηλεκτρικά ποδήλατα είναι και αυτό ένα πολύ θετικό παράδειγμα. Πρέπει να δούμε πώς θα προσφερθεί αυτό στους πολίτες αλλά και στους τουρίστες. Και για τις αερομεταφορές που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις εκπομπές. Αν είχαμε ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό θα τα είχαμε καταφέρει γιατί αυτή τη στιγμή ε, γίνονται πάρα πολλές παρακάμψεις, πάρα πολλές περιτές ε, αερομεταφορές και θα πρέπει φυσικά να ενισχυθεί και η ηλεκτρική κινητικότητα που θα τροφοδοτείτε με ηλεκτρική ενέργεια κτλ. κτλ αλλά θα μπορούσαν να συμβάλλουν όλα αυτά και στη μείωση της ηχορύπωσης. Η κυρία Κούλεν και σας παρακαλώ εσάς τους τρεις εδώ μπροστά να μιλάτε λίγο πιο σιγά. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μεγαλύτερη αλλαγή που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη αφορά την νοοτροπία των ανθρώπων. Και αυτή η αλλαγή νοοτροπίας είναι η δυσκολότερη αλλαγή από όλες. Χρειαζόμαστε διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όλων των τομέων και κλάδων. Θεωρώ ότι η διασυνοριακή συνεργασία στην Ευρώπη δεν είναι επαρκής ούτε είναι παρκής η συνεργασία εδώ εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ ε, των επιτροπών που είναι ε, υπεύθυνες για το περιβάλλον και τις μεταφορές. Δεν ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι και με αυτόν τον τρόπο σπαταλούμε πολύτιμους πόρους. Χρειαζόμαστε επίσης μεγάλα πιλωτικά έργα. που θα αφορούν τα εναλλακτικά καύσιμα, τις καινοτομίες, τα νέα οχήματα. Και το τι θα γίνει με τα παλιά οχήματα. Τι θα μπορούσε να γίνει με αυτό το retrofitting. Πώς θα μπορούσαν να επανεξοπλιστούν παλιά οχήματα ώστε να ανταποκρίνονται και στα νέα κριτήρια. Έχουμε λοιπόν χρηματοδοτικά μέσα τα οποία δεν αξιοποιούνται σωστά. Θα μπορούσε δηλαδή να ανανεωθεί και ο παλιός εξοπλισμός και αυτό αποτελεί μια ευφυή προσέγγιση περιβαλλοντική. Δεν χρειάζεται να πετα, να πετιέται στα σκουπίδια ο παλιός εξοπλισμός μπορεί κανείς και να τον ανανεώσει. Να τον αναβαθμίσει δηλαδή. Επίσης, ο ενίος ευρωπαϊκός ουρανός αντιμετωπίζει προβλήματα ακριβώ γιατί δεν, έχουμε, δεν υπάρχει συντονισμό, δεν υπάρχουν κοινέ λύσει, δεν υπάρχουν κοινέ προσεγγίσει. Άρα χρειαζόμαστε κοινές, μια κοινή προσέγγιση και ως προς την τιμολογιακή πολιτική, γιατί αυτό ενδιαφέρει τους καταναλωτές, τους πολίτες. Και οι αυξανόμενες εκπομπές που, που οφείλονται στις μεταφορές είναι μια ανησυχία που υπάρχει παγκόσμια και νομίζω ότι θα πρέπει πανευρωπαϊκά να εξευρεθεί μια ενιαία ε, προσέγγιση θα ήθελα η Ευρώπη να αποτελέσει την πρωτοπορία παγκοσμίως για την εξέβρεση λύσεων στον τομέα των μεταφορών. και στη θέσπιση μέτρων ενίσχυσης της κινητικότητας, κάτι που μάλιστα θα μπορούσε να αποτελέσει και εξαγωγικό ε, προϊόν της Ευρώπης, γιατί ανάλογα προβλήματα υπάρχουν στην Κίνα, στη ΣΥΠΑ. Και αν η Ευρώπη καταφέρει να ε, κατακτήσει ηγετική θέση, αυτό θα μπορούσε να της αποφέρει πολλαπλέον εκτήματα και παγκοσμίω. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, πρώτο και κύριο μέλημά μας θα πρέπει να είναι η αλλαγή νοοτροπίας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ η κυρία Ντέλη. Ε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και ευχαριστούμε που έχουμε και πρόσβαση σε αυτήν την έκθεση για τις μακρινές αποστάσεις. Το πρώτο τμήμα της έκθεσης προσπαθεί να δείξει ακριβώς τις δείκτε, τους δείκτες και την πρόοδο που σημειώνεται προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μάθω πώς επηρεάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως τα ε, ε, έξοδα, τις δαπάνες για τις μακρινές αποστάσεις ε, και στον αεροπορικό τομέα ποιος είναι ο αντίκτυπος του στη, στο περιβάλλον και δεν μιλάω μόνο για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αλλά πραγματικά μιλάω για το επίπεδο των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου όσον αφορά τώρα τη μείωση της συγχωρήπανσης ε, στις μεταφορές μακρινών αποστάσεων που είναι κάτι διόλου αμεληταίο. Μιλήσανε όλοι για ε, την κινητικότητα. Εγώ είμαι η συγγήτρια για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν, κατά την άποψή σας, ποια είναι τα σημαντικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν αμέσως για τη βελτίωση του περιβάλλοντος στις αστικές ζώνες. Γιατί είναι σήμερα ένα θέμα δημόσιας υγείας, υπάρχουν, ε, υπάρχει κορύφωση της ε, της ε, ε, ατμοσφαιρικής ε, μόλυνσης λόγω του δίζελ και θα ήθελα να μάθω κατά την άποψή σας πώς μπορούμε σήμερα να έχουμε μια πραγματική, ένα πραγματικό σχεδιασμό σε, στην αστική κινητικότητα, δεδομένου ότι υπάρχει επικουρικότητα και όλα τα σχετικά. Υπάρχουν πόλεις που λένε ότι κάνουμε ε, Κυριακή χωρίς αυτοκίνητα. Έχει όντως αντίκτυπο κάτι τέτοιο, έχει αποτέλεσμα. Και για τη διαχείριση της κινητικότητας, πώς γίνεται, πώς μπορούμε σήμερα να δουλέψουμε για αυτή την πράσινη ε, επιμελητία, ε, διότι υπάρχει πίσω από αυτό μια ολόκληρη σειρά θέσεων απασχόλησης που δεν είναι καθόλου αμεληταία και το είπε και συνάδελφος προηγουμένως, είναι ένα θέμα πολιτικού χειρισμού γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ε, θέματα που έχουν να κάνουν ε, με, το, με τη μεταφορά με το αυτοκίνητο. Βέβαια τώρα ε, υπάρχει τον 21ο αιώνα μία μετάβαση πέρα από τα αυτοκίνητα, στα τραμ, σε άλλου είδους μεταφορές και τι θα γίνει και με το πρόγραμμα Juncker, γιατί δεν ξέρω ακριβώς αν έχετε αναλύσει το πρόγραμμα Juncker βάσει των προγραμμάτων που έχουμε στη διάθεσή μας. Ποια είναι η άποψή σας για το πρόγραμμα Juncker σε σχέση με, το, ε, με την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ μια και μιλούμε για τις περιβαλλον... τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα, τι περιβαλλοντικές συνέπειες ε, των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων, μου φαίνεται λίγο παράδοξο το ότι δεν ε, μιλάμε για τα περιβαλλοντικά αυτοκίνητα, τα, περιβαλλοντικά φορτηγά, έτσι τα λέμε στη Σουηδία. Μπορεί κανείς ε, να μεταφέρει πολύ περισσότερα εμπορεύματα κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ έχω δουλέψει σε αυτό το τομέα. Ε, Οι 21 τόνοι χάρτου, για παράδειγμα, μπορεί να πρέπει να μεταφερθούν στη Γαλλία ε, είναι χαζό να χρησιμοποιεί κανείς πάρα πολύ μικρά ε, φορτηγά. Όταν λοιπόν μιλάμε για περιβαλλοντική διάσταση, είναι προφανώς ε, η καλύτερη λύση, η λογικότερη λύση να επιβαρύνουμε τα ε, φορτηγά με όσο το δυνατόν περισσότερα εμπορεύματα. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε το ίδιο δικό δίκτυο με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ξέρω ότι εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση για τα φορτηγά που δεν έχουν πολλές άλλες χώρες. Η Γερμανία, για παράδειγμα, σε μικρές ε, πόλεις ή μικρά χωριά δεν μπορεί να περάσουν αυτά τα τεράστια φορτηγά από το δικό δίκτυο που υπάρχει ίσως να ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 30 μέτρα, αυτοκίνητα 30 μέτρων ε, για να μπορούμε να μεταφέρουμε πολύ περισσότερους τόνους. Ε, βέβαια είναι γεγονός ότι πρέπει να γίνει μερικές φορές μεταφορά από το ένα φορτηγό στο άλλο όταν δεν μπορεί ένα πολύ μεγάλο φορτηγό να περάσει από ένα συγκεκριμένο δικό δίκτυο. Αλλά για να πάμε από το α στο β η πιο περιβαλλοντική λύση είναι να έχουμε βαρύτερα, μεγαλύτερα και μακρύτερα φορτηγά, τα οποία μπορούν να, να μεταφέρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όγκο εμπορευμάτων. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται αυτό. Προσπαθείτε να αξιοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα περισσότερα εμπορεύματα στο ίδιο φορτηγό για να μειωθεί ε, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και ατμοσφαιρική ρήπανση. Και εγώ θα ήθελα να πάρω το λόγο τελευταίος και μετά θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε για τους στόχους που αναφέρατε στην αρχή. 6% μείωση μέχρι το 2050, πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Αλλά αν δεν κάνετε το πρώτο βήμα, δεν θα φτάσουμε στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μικρότερου μεσοπρόθεσμου, ενδιάμεσου στόχου. Και νομίζω ότι στη Λευκή Βίβλο υπάρχει ένα πάρα πολύ ε, καλό παράδειγμα. Να λέμε, α πούμε, ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τους στόχους της Επιτροπής 2030 και 2050. Θέλουμε για τις μεταφορές ειδικότερα να μειωθεί ε, το επίπεδο των εκπομπών. Ποια είναι η δική σας άποψη, πώς ε, ε, οι σιδηροδρομικές μεταφορές θα επιτύχουν τους στόχους τους ή ο τομέας των, της ναυτιλίας πώς θα μπορέσει να επιτύχει τους στόχους που του αναλογούν. Δεν το αναφέρατε κι εσείς στη μελέτη σας Είπατε ότι 70% της ατμοσφαιρικής ρήπανσης προέρχεται από τις μεταφορές αστικές ζώνες. Εμάς ο Υπουργός Μεταφορών μας μας είπε ότι αυτό είναι αλήθεια. Πώς μπορούμε λοιπόν να το εξασφαλίσουμε. Τα 15 δισεκατομμύρια από το πρόγραμμα Juncker όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις οδικές μεταφορές αν δεν ασκήσουμε πιέσεις. Μήπως θα μπορούσαμε ένα τμήμα να το διαθέσουμε στο μετρό, στο τραμ, ε, στην ε, διασύνδεση μεταξύ των περιφερειών και αν όχι, για ποιο λόγο δεν το κάνουμε αυτό, γιατί αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πετύχει κανένα στόχο όσον αφορά τώρα τα φορτηγά. Προφανώς με ενδιαφέρει αυτό, είναι γεγονός ότι αλλάζει ο τρόπος θεώρησης των αυτοκινήτων και το είπατε κι εσείς ε, αναφέρατε τους στόχους που έχουν τεθεί πλέον. Ξέρουμε ότι η βιομηχανία έχει ήδη παραπονεθεί γιατί έχουν ε, ήδη επιτύχει τους στόχους δύο χρόνια πριν από την προθεσμία γιατί τα λόμπι είναι πάρα πολύ καλά σε αυτήν την, αυτοκίνητο, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Για ποιο λόγο όλα αυτά τα πράγματα δεν ε, μπορούν να γίνουν και στον τομέα των ε, εμπορευματικών μεταφορών. Για παράδειγμα μιλάω για την κυκλοφορία των φορτηγών. Είναι εκπληκτικά τα ποσοστά ε, στα ε, φόρτηγα. Δεν λέει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Είναι δυνατόν, είναι περίεργο. Ξέρετε ότι η λευκή βίβλος ε, πρέπει ίσως να αναθεωρηθεί για αυτά τα θέματα. Αν μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές από τα φορτηγά, η μακροπρόθεσμη ατμοσφαιρική ρήπανση όντως θα ε, μειωθεί για την ε, αεροπλοεία. Τεράστιος αντίκτυπος, ο αντίκτυπος της, ε, γιατί έχει τρεις-τέσσερις φορές παραπάνω συνέπειες στην ατμόσφαιρα από τις υπόλοιπες μεταφορές. Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά γι' αυτό. Πρώτον γιατί, πρώτον, επι, πρώτον γιατί επιδοτείται και είναι, ε, επιδοτείται η αεροπλοεία και αυτό δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Μιλήσατε επίσης για τα βιοκαύσιμα, μιλήσατε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν τα ηλεκτρικά οχήματα όταν ταξιδεύουν, ε, ναι μεν δεν ε, καταναλώνουν τίποτε, αλλά άμα δει κανείς τον κύκλο ζωής και τον τρόπο της ανακύκλωσής τους, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, είναι ότι ουσιαστικά ε, είναι ότι είναι πιο δύσκολη η ανακύκλωσή τους από τα κανονικά αυτοκίνητα. Μου είπε, ας πούμε, ε, ο ομοσπονδιακός μας οργανισμός ότι μπορεί να ε, μειωθεί το κόστος κατά 25% και μιλάω για το, για το τέλος του κύκλου ζωής. Αυτά λοιπόν από μένα. Περιμένω λοιπόν τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ για τις 96 ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απλουστεύσω τα πράγματα, μην απαντώντας συγχωριστά σε κάθε ερώτηση. Θα τις ομαδοποιήσω κάπως. Αν κάτι λείψει, θα μου το υπενθυμίσετε. Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αφορούσαν το αστικό περιβάλλον. Και σωστά. Απατώντας και στη γαλλική παρέμβαση, τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στα αστικό περιβάλλον. Το αστικό σύστημα θεωρείται περίπλοκο. Δεν υπάρχει σαφής λύσης. Δεν μπορούν οι σύμβουλοι να δώσουν συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος. Πολλά μέτρα εξαρτώνται από το πλαίσιο. Και μια παλιά ε, πόλη όπως η Μπρίζ εδώ ε, διαφέρει από μια σουηδική πόλη όπως η Μέα που έχει διαφορετική μορφή εξαρτάται πόλη από τις υποδομές που υπάρχουν. Το όλο δυναμικό της πόλης από την εξέλιξη της πόλης. Η ιδιαιτερότητα του πλαισίου είναι σημαντικότατη. Υπάρχουν πόλεις στην Ευρώπη που κινούνται σωστά, κινούνται προς πιο βιώσιμες ε, μεταφορές. Τα τελευταία δύο χρόνια είχα τη χαρά να ζω στην Κοπενχάγη. Πάνω από 82% των μεταφορικών μέσων της πόλης ε, είναι τα ποδήλατα 42% και 40% δημόσιες μεταφορές ή με τα πόδια. Υπάρχει ένα σύστημα δρόμων, ποδηλατοδρόμων όταν χιονίζει στην Κοπενχάγη πρώτα καθαρίζουν τους ποδηλατόδρομους. Υπάρχει οργάνωση, υπάρχουν επιχειρήσεις. Είναι σύνηθε ο διευθυντής και υπάλληλοι σε μια εταιρεία να καταφθάνουν με ποδήλατο, να έχουν χώρο να σταθμίσουν το ποδήλατο, να μπορούν να κάνουν τον ντου τους μετά. Υπάρχει διασύνδεση με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Υπάρχουν αυτοκίνητα στην πόλη, κινούνται διαφορετικά όμως. Είναι πλήρες το σύστημα. Αν δείτε τι δημόσιε μεταφορέ και το ρόλο που παίζουν. Υπάρχουν διαφορετικά παραδείγματα στην Ευρώπη πιθανότατα να γίνονται παρόμοιες επενδύσεις στις δημόσιες μεταφορές, αλλά με ποικίλα αποτελέσματα. Είναι και θέμα σχεδιασμού των συστημάτων με το βέλτιστο τρόπο. Να έχουμε τεχνική συγκοινωνία, υψηλής ποιότητας, ασφαλή συγκοινωνία, ούτως ώστε ο κόσμος να το χρησιμοποιεί το σύστημα. Από την εμπειρία μου πιστεύω ότι η Κοπενχάγη είναι ένα άριστο παράδειγμα ε, κάτω από το κοινοβούλιο εδώ έχετε ένα υπέροχο σταθμό. Αν θέλετε να φτάσετε όμω στο αεροδρόμιο, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι απίστευτο να σχεδιαστεί κάτι όπως σχεδιάστηκε. Στο αστικό περιβάλλον λοιπόν. Είναι περίπλοκο το σύστημα το αστικό. Μετά ξέρουμε ποιος είναι αντίκτυπος των οχημάτων, των αυτοκινήτων με ε, διζελοκινητήρες. Ο αντίκτυπος είναι πολύ μεγάλο στο αστικό περιβάλλον πρέπει να εξετάσουμε και τι προωθεί τα αντιζελοκίνητα αυτοκίνητα για ιδιωτική χρήση σε χώρες. Ε, χρειάζεται ευνοϊκή φορολόγηση για τα καύσιμα και τα αυτοκίνητα για να προωθήσει κανείς τους κινητήρες δίζελ. Περιβαλλοντικές επιδοτήσεις αφορά και συνήθειες. Από τη δική μου εμπειρία σε αυτή τη χώρα, ένα αυτοκίνητο με δίζελ είναι εύκολο να αγοραστεί. Να αναφερθώ και σε άλλα θέματα. Η τιμολόγηση και οι σχετικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται εν γέννη στα συστήματα κινητικότητας και μεταφορών έχει τεράστια επιρροή στα αποτελέσματα. Ξέρουμε το Λονδίνο με το σύστημα τιμολόγησης. Αν μειωθεί ο αριθμός των αυτοκινήτων στην πόλη κάποια στιγμή έχει τεράστιο αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης στην πόλη και στις κινήσεις. Αν εφάρμοζες τιμολόγηση με πιο ευφυή τρόπο θα μπορούσες να επηρεάσει και τη ζήτηση της κινητικότητας και των μεταφορών και την κατανομή κατά τη διάρκεια της ημέρας και το πότε και πού χρησιμοποιεί ο κόσμος τα μέσα μεταφορών. Αν υπάρχει ποικίλη ε, προσέγγιση σε κάθε γειτονιά, περιπλέκονται τα πράγματα. Άρα χρειάζεται συντονισμός και σε διασυνοριακό επίπεδο. Η διασυνοριακή πτυχή. Τη θίξατε αρκετή από σας. Ωστόσο δώσω ένα παράδειγμα. Αναφέρθηκα στην Κοπεχάγη. Την έβαλα σαν καλό παράδειγμα. Απέχει μόνο 900 χιλιόμετρα από εδώ. Αν θέλω να πάω εκεί σιδηροδρομικά, πρέπει να πάρω και την πιτζάμα μου. Αξιοσημείωτο αυτό. Ξέρω ότι ετοιμάζουν μια σύραγγα που θα διευκολύνει τα πράγματα. Αλλά η κατασκευή διασυνοριακών υποδομών που επιτρέπει στον κόσμο να κάνει επιλογές, να μην υποχρεώνεται να πάρει κάποια μέσα να κάνει επιλογές, είναι κάτι που απαιτεί σαφής κατευθύνσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θέλουμε να το πετύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, αν ισχύει το βασικό σχέδιο για την Ευρώπη μόνο στις μεταφορές, όχι, το master plan, δεν νομίζω. Ισχύει και για τις υποδομές, διασυνδέσεις που δεν λειτουργούν, δεν υφίστανται. Και θέλουμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις. Κάποιοι είπαν κατά πόσο μπορούμε να είμαστε πιο αποδοτικοί όσον αφορά το πώς κινούμεθα, όσον αφορά τα μεγάλα φορτηγά ή τους ε, διαδρόμους που χρησιμοποιούν τα αεροσκάπη στις υπερπτήσεις. Είναι κάτι που το εξετάσαμε και σε αυτή και σε άλλες εκθέσεις. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα. Αν θέλουμε να μειώσουμε κατά 60% πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα και άμεσα. Δύο είναι σημαντικά. Πρώτον, να αποφύγουμε επενδύσεις σε πράγματα που μας παγιδεύουν και μας οδηγούν σε μακροπρόθεσμη μη βιωσιμότητα. Θέλουμε, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους του 2030 ποικιλοτρόπως, εστιαζόμενοι και διαθέτοντας οικονομικούς πόρους, έρευνα και τεχνολογία σε πόρους που θα μας οδηγήσουν στους στόχους του 2020 και του 2030 αλλά που θα παγιδεύσουν κεφάλαια στα παλιά συστήματα και θα μπορούσαν να εμποδίσουν να επενδύσει κανείς τη μετάβαση προς το 2050. Οι θεσπίζοντες την πολιτική μαζί με τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να εξασφαλίσουν το ότι οι πραγματοποιούμενες επενδύσεις όχι μόνο οδηγούν ε, σε επενδύσεις σε κλειδωμένα συστήματα, αλλά ανοίγουν και διαδρόμους για μελλοντικούς στόχους. Και οι δύο τομείς δεν ταιριάζουν πάντα. Um, when we are Όταν μιλάμε για εναλλακτικά καύσιμα και τα σχετικά αυτοκίνητα, που σχετίζεται με αυτό που αναφέρατε, ποια τρένα ρηπαίνουν περισσότερο, εξαρτάται και από τα καύσιμα. Ο ποικίλει. Αν παράγεις την ηλεκτρική ενέργεια των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με εγκαταστάσεις που παράγουν ε, πολλά αέρια του θερμοκηπίου και ρηπαίνουν δεν κερδίζει πολλά. Ο ηλεκτρισμός που χρησιμοποιείται από τα τρένα εξαρτάται από την πηγή του ηλεκτρισμού ή συνέπεια όσον αφορά ε, το δεξιού άνθρακος. Σε τοπική ρήπανση είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά μιλάμε για γενικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Έχουμε ετοιμάσει εκθέσεις επίσης για έμεσες αλλαγές χρήσεως της γης και αντίκτυπο των βιοκαυσίμων. Και συμπεράναμε ότι πράγματι τα βιοκαύσιμα μπορούν να συμβάλλουν στη λύση. Αλλά αν δεν κινηθεί σωστά υπάρχουν τεράστια συν και πλήν. Χρειάζεται λοιπόν προσεκτική ανάλυση των επιλογών. When it comes Στον για την Ευρώπη και ποια τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να προχωρήσει. Κέρδης, αποδοτικότητα σε μέγεθος και να πω στον κύριο Λούντγκρεν εδώ ότι υπάρχουν και πιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι και άλλη προσέγγιση μέσω μειώσεω των μεγεθών σε αστικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια κέρδη αποδοτικότητα αν κινηθεί διαφορετικά. Αφορά και τα δύο άκρα του φάσματος που μπορούν να εξεταστούν. Ίσως σε εκπλήσει, αλλά 25% της έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη πηγαίνει στην αυτοκίνητη και στις μεταφορές 25%. Τεράστιο ποσό, τεράστιο. Λοιπόν, επενδύουμε. Τεράστια ποσά. Ιδιωτικού και δημοσίου κεφαλαίου για έρευνα στον τομέα των μεταφορών. Η πρόκληση για την Ευρώπη είναι να το κάνει αυτό υπό το φως των μακροπρόθεσμων στόχων. Να σας υπενθυμίσω και κάτι και σαν περιβαλλοντική υπηρεσία το ξέρουμε άριστα ότι το 7ο πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το περιβάλλον έχει ένα όραμα για το 2050 για μια οικονομία χαμηλού άνθρακος. Μια κυκλική πράσινη οικονομία και οικοσύστημα παντέχει. Η επιλογή που θα γίνει όσον αφορά τι μεταφορέ και την κινητικότητα είναι κρισίμου σημασία για την επίτευξη των στόχων. Μετά, όταν επενδύει κανείς στον τομέα μεταφορών και κινητικότητας στα σχετικά συστήματα, είναι να χρησιμοποιείς διάφορους ε, πύχης και μέτρα για να μπορείς να κρίνεις τις πολιτικές και τις επενδύσεις που έχουν στόχο τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα. Χρησιμοποιούνται με αυτή την προσέγγιση, ε, βελτιώνουμε την αποδοτικότητα μπορείς έτσι να κρίνεις τις δημόσιες δαπάνες βάσει του προγράμματος Juncker ή σε επίπεδο κράτους μέλους. Δεν θέλω να προβώ σε πολιτικές δηλώσεις. Όσον αφορά το πρόγραμμα πολιτικής, δεν είναι ο ρόλος του φορέα μας αυτός. Οι εκθέσεις μας και τα στοιχεία δείχνουν σαφώς πού πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά οι επενδύσεις. Δύο-τρεις αναφέρθηκαν στο θόρυβο. Ετοιμάσαμε την πρώτη έκθεση περιθορύβου το Δεκέμβριο. Εξεδόθη. Δύσκολο θέμα. Τα στοιχεία λείπουν. Η ποιότητά τους δεν είναι άριστη. Ξέρουμε ότι κυρίως αστικές περιοχές ο θόρυβος και η κυκλοφορία είναι αλληλένδετα και μπορεί κανείς να κάνει σαφείς επιλογές όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και στους δρόμους και στα οχήματα και διάφορους τείχους μπορεί να κατασκευάσει για να προστατεύει τα σπίτια από τον ήχο και η χωροταξία είναι μια άλλη διάσταση. Η ζήτηση για τις μεταφορές ξεκινά από την χωροταξική κατανομή των κοινωνικών δραστηριοτήτων. Πολλά μπορούν να γίνουν εκεί. Εναέρια κυκλοφορία. Πολύ το αναφέρατε αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα απ' όλα αυτό είναι θέμα διεθνές, να μην πω παγκόσμιο. Όλοι γνωρίζετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα, ότι είναι δύσκολο θέμα, δύσκολο να συζητηθεί. Όσον αφορά τη διατλαντική συζήτηση, και τις χώρες ανάπτυξης, με τις χώρες BRICS, τις χώρες μεσαίου εισοδήματος. Ποια είναι η προσδοκία ότι οι αερομεταφορές τις επόμενες δεκαετίες, αν δεν αλλάξει τίποτα, ε, θα αυξηθούν πολύ, τρεις φορές με τέσσερις φορές. Άρα, αν δεν αλλάξουμε το πώς επηρεάζουν οι αερομεταφορές το κλίμα, αλλά και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα πράγματα θα γίνουν αρκετά δύσκολα. Δύσκολα για να πετύχουμε τους στόχους που έχει θέσει η Ευρώπη και ο κόσμος όσον αφορά τη μείωση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. αερίου του θερμοκηπίου. Το ίδιο ισχύει και για την αυσιπλοεία. Σε μεγάλο βαθμό έχουμε αρκετά παλιά τεχνολογία που χρησιμοποιείται, βελτιώνεται η απόδοσή τους με την πάρο των ετών, αλλά νέα τεχνολογίες θα κάνουν τη διαφορά. Και οι πιο καινοτόμε επιχειρήσει στην αυσιπλοεία της Ευρώπης πειραματίζονται με νέες τεχνολογίες για τους κινητήρες των μεγάλων πλοίων. Άρα υπάρχουν θέματα να εξεταστούν. Λοιπόν, Τέλος, κάποιοι αναφέρατε ότι είναι σχεδόν αξίωμα ότι η ζήτηση για μεταφορές θα αυξηθεί. Δεν θα ήταν συνετό βάσει της ανάλυσής μας να θεωρήσουμε δεδομένη τη ζήτηση και να εστιαστούμε επί της προσφοράς και των υποδομών Υπάρχουν πιστικές μελέτες που δείχνουν ότι ένα απλό καταναλωτικό αγαθό όπως μετακινείται από χώρα σε χώρα εντός χωρών, εντός Ευρώπης και αν δει κανεί εξωτερικές πτυχές της κινητικότητας βλέπει ότι είναι τεράστιος αντίκτυπος. Αν εξετάσουμε παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και ευρωπαϊκές παρεμφερείς και πώς παράγονται οι ροές της κινητικότητας και η τιμολόγηση, θα δείτε υπάρχουν προβλήματα. Θα μας πούνε τι θέλετε να βγάλουμε εκτός σημαντικό τμήμα της οικονομίας. Υπάρχουν πιστικές μελέτες που δείχνουν ότι μπορείς να έχεις και άλλους τρόπους οργανώσεως κινητικότητας που να, παράγεται να παράγονται θέσεις απασχόλησης, λιγότερες εξωτερικές συνέπειες, λιγότερο κόστος για τα συστήματα υγείας και τα άλλα συστήματα. Και το τελικό καθαρό αποτέλεσμα για την οικονομία είναι θετικό. Και δημιουργείς ποιοτικές θέσεις απασχόλησης με θετική επιρροή για την κοινωνία. Χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση και σε συνάρτηση με τους μακροπρόθεσμους στόχους. Θα σταματήσω εδώ. Λυσμόνησα κάποιες λεπτομέρειες. Α, εκπομπές φορτηγών. Δεν διαμορφώνουμε πολιτική. Αξιολογούμε πολιτικές. Ξέρουμε ότι λείπουν οι στόχοι για μεταφορές περιβάλλον και άλλα θέματα είδαμε ότι οι πολιτικές τείνουν να έχουν θετικές συνέπειες όταν έχουν στόχους, όταν είναι φιλόδοξες πολιτικές, όταν σωστά διατυπωμένες και σωστά εφαρμοσμένες. Οι σαφείς στόχοι είναι βασική συνιστόσα πολιτικών που καταλήγουν σε σαφή αποτελέσματα. Και να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό στις σημερινές πολιτικές και το κλίμα. Σε τρία επίπεδα επιτυχάνονται αποτελέσματα. Περιβαλλοντικός αντίκτυπος αντίκτυπος για την υγεία, αντίκτυπος για, για καινοτομία, εφευρέσεις, πνευματικά δικαιώματα. Είναι ο τομέας των οικολογικών προϊόντων που από την κρίση ανέβηκε στα 4 εκατομμύρια θέσει απασχόληση. Υπάρχουν διπλώματα ευρεσιτεχνία περισσότερα στον τομέα προστασία του περιβάλλοντο από το 2008 μέχρι σήμερα από ό,τι ποτέ. Υπάρχει εξαγωγική ζήτηση, γίνονται εξαγωγέ από την Ευρώπη, αλλά υπάρχουν ωφέλη και στα τρία επίπεδα. Και είναι σημαντικά για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Μπρόινιγκς για την παρουσία σας ήταν εξαιρετική, μας δίνει επιχειρήματα. Δεν είστε βεβαίως φορέας ε, χάραξης πολιτικής, αλλά σας διαβεβαιώ ήταν εδώ και η Κομισιόν, σας άκουσε, οπότε όταν θέτουμε εμείς τα ερωτήματα θα, ε, για το πού κατευθύνονται τα χρήματα θα ξέρουμε πώς μπορούμε να ε, επιτύχουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και φυσικά θα συνεχίσουμε ε, τη συνεργασία μας. Άκουσα ότι ο κύριος Μπράουνινγκ θέλει να κάνει μια παρατήρηση, αλλά τον σταματήσατε με την ε, ερώτηση σας για, τους ε, για τα φορτηγά. Την επόμενη φορά θα πρότεινα η παρουσίαση να διαρκέσει δύο ώρες. Θα το κάνω αυτό, λέει ο πρόεδρος. Ευχαρίστως και το γεγονός ότι η πρόταση μάλιστα ε, υποβάλλεται από εσά είναι ακόμη καλύτερο. Το είχα σκεφτεί και εγώ, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε την επόμενη φορά. Κύριε Μπρόνιξ, να έρθετε δύο ώρες και τώρα θέλει να απαντήσει. Γιατί φυσικά αν θέλουμε να του δώσουμε δύο ώρες μπορούμε σήμερα να του δώσουμε ένα λεπτό. Θέλω απλά να πω ότι αν έχετε πιο λεπτομερείς ε, ερωτήσεις για τις εκθέσεις μας για τις μεταφορές και το περιβάλλον μπορείτε βεβαίως να απευθυνθείτε στον οργανισμό μας. Θα σας απαντήσουμε εντός των ε, προβλεπόμενων ωραίων, ε, ε, και θα σας παράσχουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας, τις γνώσεις μας για τα θέματα που θα μας θέσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το 18, έλεγχος των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας. Καλωσορίζω τον κύριο Ονίδη από την Γενική Διεύθυνση MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Και εδώ οι τρεις σας, σας παρακαλώ λίγο πιο ήσυχα ή αλλιώς βγείτε έξω από την αίθουσα γιατί δεν γίνεται. Τώρα φταίνει η άλλη. Έχετε δίκιο μάλλον. Thank you. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Η ασφάλεια είναι σημαντικότατο ζήτημα πράγματι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Έχουμε ένα νέο τομέα δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια νέα αρμοδιότητα που ανατέθηκε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Κάποιες νέες αρμοδιότητες που βασίζονται σε ένα ε, χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί μιλάμε για έναν κανονισμό και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Πρόκειται για νομοθεσία που συμπληρώνεται και επικαιροποιείται διαρκώς μέσω εκτελεστικών πράξεων στις οποίες συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο παρατηρήσεις και στη συνέχεια θα δώσω τον ε, λόγο στον Κάλλος Μέστρε για να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι ο κανονισμός έχει αποδείξει ότι είναι ευέλικτος ως προς την προσαρμογή του στις ε, ε, συνθήκες που αλλάζουν και αυτές οι συνθήκες πράγματι αλλάζουν πολύ γρήγορα. Έχουμε δείξει ότι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου νομοθετήματος έχουμε εξασφαλίσει την ασφάλεια των επιβατών και μάλιστα με ε, εύλογο κόστος που ήταν μια σημαντική διάσταση που λάβαμε, ε, που λάβαμε υπόψη μας το Κοινοβούλιο στο πέρας των χρόνων έχει συνεισφέρει σημαντικότατα, αφενός γιατί μας έθετε διαρκώς το ερώτημα της αναλογικότητας των μέτρων που λαμβάνονται, να εξασφαλίζουμε δηλαδή ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι απολύτως αναγκαία και αναλογικά ως προς τον κίνδυνο που έχει αναλυθεί. Επίσης υπήρξε επικέντρωση από την πλευρά του ε, Κοινοβουλίου στην προώθηση των νέων τεχνολογιών για την απλούστευση και την μείωση των, του κόστους των ε, μέτρων ασφαλείας και τέλος μας υπενθύμιζε πάντοτε ότι πρέπει να έχουμε κάνος, κανόνες που θα πρέπει να είναι απλοί ώστε να μπορεί κανείς να τους εξηγήσει στους επιβάτες αλλά να μπορούν και οι εθνικές αρχές να τους εφαρμόζουν. Και Υπάρχει και ο διεθνής ε, τομέας δραστηριοτήτων. Σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα με τις ΙΠΑ, έχει υπάρξει ένας βαθμός ολοκλήρωσης, ενσωμάτωσης. Πολλοί από εσά επισκέφθηκαν την Ουάσιγκτον την προηγούμενη εβδομάδα και είδατε κι εσείς ότι ο βαθμός ολοκλήρωσης ε, συνεργασίας και αμοιβαίας αναγνώρισης των κανόνων που ισχύουν στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχει προχωρήσει και αυτό δεν αφορά μόνο τις ε, ΗΠΑ αλλά και άλλους εταίρους, την Αυστραλία, τον Καναδά και όλο ένα και περισσότερο ε, και άλλες χώρες από ολόκληρο τον κόσμο που χρειάζονται τη δική μας βοήθεια, τη δική μας αρρωγή προκειμένου να θεσπίσουν καλύτερους κανόνες ασφαλείας που δεν θα ισχύουν μόνο για τις επιβατικές μεταφορές αλλά και για τις εμπορευματικές μεταφορές και μάλιστα ε, από ορισμένες απόψεις ε, είναι πιο σημαντική η θέσπιση τέτοιων κανόνων στις εμπορευματικές μεταφορές γιατί έχουμε κοινούς κανόνες. Και δίνω τώρα τον λόγο στον Κάρλος για να μας παρουσιάσει το πλαίσιο που ισχύει σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Θα διατρέξω κάποιες διαφάνειες σας. Έχω μια παρουσίαση. Αν τα καταφέρω. make time for Πολύ γρήγορα για να έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις. Θα σας παρουσιάσω τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε στην ασφάλεια της αεροπορίας. Αυτό που χρειάζεται να σας πω αρχικά είναι ποιοι είναι οι στόχοι που έχουμε θέσει. Πρώτος στόχος είναι η προστασία ε, της πολιτικής αεροπορίας έναντι παράνομων παρεμβάσεων. Δηλαδή κατευθυντήριες οδηγίες και αυτό συνδέεται με, τις, ε, με τα πρότυπα ασφαλείας του ΙΚΑΟ όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια. Στόχος είναι η θέσπιση κοινών κανόνων που θα εφαρμόζονται από όλα τα κράτη-μέλη με έναν τρόπο που θα μπορεί και να ελέγχεται από τις ε, κατάλληλες αρχές των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημαντικό είναι ότι αυτό το σύνολο κανόνων είναι πιο ε, αυστηρό από, τους, από τα πρότυπα του ΙΚΑΟ. Απαιτείται συντονισμός που είναι ένας από τους θεμέλους λίθους του συστήματός μας. Σημαίνει επίσης ότι η συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σημαίνει ε, αυτόματη συμμόρφωση με τα, με τα πρότυπα του ΙΚΑΟ. Ε, το η βασική δομή του συστήματός μας βασίζεται στην νομοθεσία πλαίσιο, τον κανονισμό 300 του 2008, που αποτελεί το βασικό κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που συμπληρώνεται από ε, εκτελεστικές κατευθυντικές πράξεις. Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας είναι δημόσιο, υπάρχει και μία απόφαση που έχει έναν ε, βαθμό εμπιστευτικότητας. Αυτή είναι η βασική νομική δομή που ισχύει και έτσι εφαρμόζουμε τα στοιχεία. Βλέπετε ότι ο κανονισμός πλαίσιο προβλέπει τις βασικές αρχές αυτού του συστήματος όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, το ποια είναι αυτά τα βασικά πρότυπα που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εργαλεία που απαιτούνται σε εθνικό επίπεδο, Υπάρχουν και οι έλεγχοι, επιθεωρήσεις, αλλά και η αναγνώριση στοιχείων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του συστήματος. Το γεγονός ότι έχουμε αυτούς τους κοινού κανόνες σε όλα τα 28 κράτη-μέλη και τα μέλη του ΕΟΧ μπορούμε να ε, εξασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια. Γιατί αυτό μας ε, δίνει ε, τη δυνατότητα καλύτερης επιχειρησιακής ε, ε, ετοιμότητας και εξοικονόμησης πόρων γιατί υπάρχει μόνο ένας έλεγχος στο αεροδρόμιο εισόδου. Δεν υπάρχουν άλλοι έλεγχοι σε μετέπειτα αεροδρόμια που μπορεί να πάει κανείς και αυτό εξοικονομεί τεράστιους πόρους. Οι κανόνες επίσης συμπληρώνονται από συμπληρωματικές πράξεις. Βασικότερη είναι ο κανονισμός 272 του 2009 που ε, δίνει ορισμένες λεπτομέρειες ε, και ορισμένα περισσότερα στοιχεία. Για να σας δώσω μια εικόνα. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου και εξέτασης. Και εκτελεστικές πράξεις θα ορίσουν πώς ακριβώς θα εφαρμόζονται αυτές οι μέθοδοι. Άρα, ο κανονισμός πλαίσιο και οι συμπληρωματικές πράξεις θα ορίσουν για ποιο λόγο θα πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένε δράσεις, με ποιον τρόπο οι εκτελεστικές πράξεις στη συνέχεια θα περιγράφουν πώς θα γίνεται όλο αυτό. Υπάρχει μεγάλο μέρος του κανονισμού που μεταφέρθηκε και στην απόφαση γιατί υπάρχουν ε, και ορισμένες, ορισμένα ζητήματα εμπιστευτικότητας. Βασιστήκαμε στις εργασίες της Επιτροπής για την ε, ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας που εργάζεται από το 2011 για την σύνταξη εκ τελεστικών πράξεων. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα που αναφέρονται στην απόφαση, την ε, επικαιροποίηση των καταλόγων των εισερχόμενων ε, εμπορευμάτων ε, δια αέρος. Υπάρχουν και κάποιες περιοδικές ασκήσεις στις οποίες εμπλέκονται και οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να μας δίνουν τα δικά τους στοιχεία για να μπορούμε να ε, τους διευκολύνουμε. Και αυτό είναι από τα σημαντικά στοιχεία. Ο κανονισμός προβλέπει την ε, Συμβουλευτική Επιτροπή των Εμπλεκομένων Φορέων που έχει συμβουλευτικό ρόλο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων όπου μπορεί να συμμετέχει ε, κάθε οργανισμός που σχετίζεται με την πολιτική αεροπορία. Έχουμε αεροδρόμια, μεταφορείς, ε, αεροπορικές εταιρείες, ε, κατασκευαστές εξοπλισμού, πιλότους. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά από που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα και μπορούν να συνδιαμορφώνουν ε, την εξέλιξη αυτών των κανονισμών και των κανόνων. Αυτό το ΣΑΓΑΣ όπως ονομάζεται, ε, έχει συμβουλευτικό ρόλο προς την Κομισιόν, ε, παρέχει εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη στην ασφάλεια της αεροπορίας και από πρακτικής άποψης προσπαθεί να ευθυγραμμίσει το έργο της Επιτροπής ΑΦΕ και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να ε, διασφαλίσουμε ότι δίνουμε αποτελεσματικές απαντήσεις στη βάση των σχολείων και των στοιχείων που μας δίνουν οι εμπλεκόμενοι φορείς όσον αφορά, μπορούν όμως και εκείνοι να θέσουν ορισμένες δικές τους προτεραιότητες ή και θέματα για περαιτέρω συζήτηση σε αυτήν την Επιτροπή. Επίσης σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι το σύστημα αυτό βασίζεται στην πραγματικότητα σε μια αρχή βασισμένη στον κίνδυνο. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, οι κανόνες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κινδύνους, στους δυνητικούς κινδύνους και να υπάρχει διαχείριση του κινδύνου. Ένα σύστημα αντιθέτως που θα ε, βασιζόταν στην αποφυγή των κινδύνων θα οδηγούσε σε τερματισμό των ροών και των μεταφορών. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα απέδιδε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει μια πολύ σαφή μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου που, διεξάγονται, που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και υπάρχει συντονισμός όχι μόνο μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής, όπως για παράδειγμα με την Γενική Διεύθυνση Home, εσωτερικών υποθέσεων, αλλά συνεργαζόμαστε και με τις εθνικές υπηρεσίε ε, και του τους φορεί που συμμετέχουν στην Επιτροπή ΑΦΣΕΚ. Στη συνέχεια οδηγούμαστε σε μια ανάλυση για το ποια είναι, ε, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιε είναι οι απειλές και στη συνέχεια αποφασίζουμε για το τι μέτρα θα ληφθούν. Και αυτά τα μέτρα πρέπει πάντοτε να είναι βιώσιμα. Δεν μπορούμε να ε, αντιδρούμε υπερβολικά ούτε μέσα σε πάρα πολύ ε, σύντομο χρονικό διάστημα αλλά πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους που είναι πραγματικά υπαρκτοί που είναι δομικοί και τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με βιώσιμο τρόπο. Έχουμε ε, επιτελέσει έργο ε, τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τους ελέγχους των επιβοτών και τους ε, κινδύνους που θέτουν, που δημιουργούν οι εκρηκτικές συσκευές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, της αξιολόγησης που κάνουμε όσον αφορά τον έλεγχο των επιβατών. Αποτελεί σημαντικό σημείο της διαδικασίας να εξασφαλιστεί ότι ο επιβάτης θα έχει μια θετική εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται και η ασφάλεια της όλης διαδικασίας. Και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, αναλογικό και αποτελεσματικό σύνολο κανόνων ώστε να εντοπίζονται οι πραγματικοί κίνδυνοι. Είχαμε κάποια παραδείγματα τα τελευταία χρόνια, τα υγρά που απαγορεύτηκαν ε, στις χειραποσκευές και το έργο που έχει γίνει Έκτοτε, για την άρση των περιορισμών μέσω της χρήσης ε, εξοπλισμού ελέγχου. Έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο και πλέον υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρει κανείς μαζί του στη χειραποσκευή του υγρά ε, από τα καταστήματα αφορολογήτων και ελπίζουμε ε, να υπάρξει οριστική άρση αυτής της απαγόρευσης υγρών μέσω του ελέγχου των υγρών. Άλλο παράδειγμα είναι ε, ο, ε, η απειλή που ε, συνιστούν οι μη μεταλλικές εκρηκτικές συσκευές. Φέτος θα προσθεθούν κάποια μέτρα ασφάλειας προκειμένου να εντοπίζονται οι συγκεκριμένες απειλές. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να τονίσουμε είναι το γεγονός ότι δεν περιγράφουμε με σαφήνεια τις μεθόδους που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αυτό που ε, παρέχουμε εμείς είναι ένας συνδυασμός μεθόδων. Τα αεροδρόμια ε, και οι εθνικές αρχές θα αποφασίζουν ποιες μεθόδους θα χρησιμοποιούν. Θέλουμε δηλαδή να δίνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Άλλο παράδειγμα του έργου που έχει γίνει αφορά τις εμπορευματικέ μεταφορές. Το 2010 υπήρξε ένα φορτίο με εκρηκτικά μέσα σε εκτυπωτή και αποτέλεσε πραγματική απειλή. Από το 2010 προσπαθήσαμε και εξασφαλίσαμε να υπάρξει ένα σύστημα για τις εισαγωγές εμπορευμάτων ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από ε, ασφαλείς πηγές. Υπάρχει λοιπόν το σύστημα ACC3 που ορίζει ότι κάθε εμπόρευμα θα πρέπει να έχει ε, διαπιστευτεί, θα πρέπει να έχει επαληθευτεί ότι κάθε εμπόρευμα έχει, προέρχεται από ασφαλή πηγή. Χρειάζεται να ε, αρχίσουμε και ένα διάλογο με τους εταίρους μας σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου αυτοί οι κανόνες που ισχύουν σε ευρωπαϊκή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνάδουν με τους κανόνες που ισχύουν παγκοσμίω και θα ε, συμπληρώνονται και θα υποβοηθούνται και από τεχνολογικά έργα που υποστηρίζουμε σε όλο τον κόσμο. Τρίτο στοιχείο είναι η τεχνολογία. Όπως ανέφερα νωρίτερα, η νομοθεσία ε, προσφέρει μια εργαλειοθήκη μεθόδων και λύσεων. Και εμείς ποτέ δεν ε, ορίζουμε συγκεκριμένες ε, τεχνολογίες που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων απειλών. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ε, ε, της διευκόλυνσης της, και, και, και, των οικονομικών διαστάσεων της λειτουργίας των αεροδρομίων. Υπάρχει και ένας κανονισμός, τον οποίο έχουμε εκδώσει, και η Κομισιόν ενθαρρύνει και την χρήση καινοτόμων έργων όπως το ACBS, το Advanced Cabin Baggage System, που, δίνουν, που διευκολύνουν και τους ε, επιβάτες ώστε να μπορούν για παράδειγμα να έχουν στη χειραποσκευή τους λάπτοπ ε, ή και κάποια υγρά. Άλλο σημαντικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας είναι η διεθνής διάσταση. Όπως είπα νωρίτερα, ο κανονισμός περιέχει ήδη, προβλέπει ήδη την δυνατότητα αναγνώρισης ε, προτύπων που ε, εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και με αυτόν τον τρόπο να επεκτείνουμε την λογική του one-stop security σε άλλα μέρη του κόσμου και μια από τις βασικές επιτυχίες μας είναι η αμοιβαία αναγνώριση προτύπων για τις εμπορευματικές μεταφορές και τις ε, εμπορευματικές μεταφορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ΕΥΠΑ. και μάλιστα ε, λαμβάνουμε μέτρα ώστε να επεκτείνουμε ακόμη περισσότερα τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος. Επίσης, Θέλουμε να επεκτείνουμε αυτές τις αρχές της αμοιβές αναγνώρισης και του One Stop Security και με άλλες χώρες. Έχουμε προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στις συζητήσεις μας με τον Καναδά, αλλά και με άλλες χώρες. Ιδιαίτερα από περιφέρειες ή όπου έχουμε ε, ενδείξεις ότι επιτελούν τεράστιο έργο όσον αφορά την εφαρμογή των προ, προ, προτύπων. Επίσης συνεργαζόμαστε με τον ΙΚΑΟ, ιδιαίτερα όσον αφορά την αρρωγή που παρέχεται σε τρίτες χώρες, προκειμένου εκείνες να ενισχύουν τα πρότυπά τους και μια ομαλή ε, ε, εφαρμογή των κανόνων ACC3 που ανέφερα νωρίτερα. Και να τελειώσω με το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα επισημαίνω ίσως τα πιο σημαντικά στοιχεία. Θα συνεχίσουμε τη θέσπιση μέτρων στη βάση της αρχής ε, που θα βασίζεται στον κίνδυνο, αποτελεί το θεμέλιο λίθο του συστήματός μας. προκειμένου να καταστούν όσο δυνατόν αποτελεσματικότητα και οικονομικά αποδοτικά. Θέλουμε επίσης να συνεχίσουμε την, ε, ε, ε, το έργο για την άρση των απαγορεύσεων μέσω της νέας τεχνολογίας και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε την θετική εμπειρία των επιβατών να μην δηλαδή δημιουργήσουμε από την άλλη πλευρά μεγάλες ουρές στον έλεγχο των χειραποσκευών. Επίσης, θα συνεχίσουμε το έργο ε, όσον αφορά το, την τεχνολογία, το One Stop Security. Η τεχνολογία εξακολουθεί να είναι μία από τις ε, προτεραιότητές μας. Θα έχουμε αυτό το ενισχυμένο, το προωθημένο σύστημα ε, χείρα αποσκευών και τέλος η Κομισιόν προετοιμάζει μία στρατηγική για την αεροπορία που θα περιέχει και ένα κεφάλαιο που θα αφορά συγκεκριμένα την ασφάλεια της αεροπορίας. Τελειώνω εδώ την παρουσίαση μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Βιμ Φαντεκάμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Τζόρτζ Μπαχ θα ήθελα να πάρει το λόγο. Εμείς είχαμε το προνόμιο να πάμε στι Ηνωμένε Πολιτείε και εσείς και εγώ και να συζητήσουμε με τον οργανισμό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των μεταφορών. Και μου έκανε εντύπωση ότι 60.000 άτομα εργάζονταν σε αυτό το τομέα, στον τομέα της ε, ε, αεροπορικής ασφάλειας. Πραγματικά είναι τεράστιος ο κλάδος και αυτό, αυτή η επίσκεψη μου δημιούργησε τις εξής ερωτήσεις. Ξέρουμε ότι 90% των επιβατών δεν είναι τρομοκράτες, θέλουν απλώς να ταξιδέψουν το όσο το δυνατόν ταχύτερα. Υπήρχαν πάρα πολλοί έλεγχοι και αυτό το γενικό πρόγραμμα τόσο διεξοδικών ελέγχων ε, ε αναρωτιέμαι αν υπάρχει περίπτωση να το έχουμε και στην Ευρώπη. Ισμαήλ Ερτούκ. Να ευχαριστήσω εκ μέρους των σοσιαλιστών την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτές οι νέες τεχνολογίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες γιατί μπορούν πραγματικά να διευκολύνουν τα ταξίδια χωρίς ταυτόχρονα να μειώνεται το επίπεδο ασφάλειας. Θα ήθελα να ε, μας δώσετε κάποιες ε, περισσότερες ε, πληροφορίες για αυτό το Advanced Baggage System Νομίζω ότι ε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το σύστημα και για τους πολίτες γιατί μπορούν μέσω αυτού να ε, διαπιστώσουν και οι πολίτες τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την διευκόλυνση και της καθημερινής τους ζωής. Αυτό και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση σας. Ευχαριστώ η Τζάκι Φώστερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Όπω είπαν και οι συνάδελφοι, ξέρετε ότι είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα στι ΗΠΑ και είδαμε όλου του αρμόδιου φορεί. Ήταν πάρα πολύ παραγωγικό, ήταν πάρα πολύ καλή η ενημέρωση που είχαμε. Εγώ ήμουν η αρχική εισηγήτρια για του ε, κανόνε των αεροδρομίων και ήταν δική μου ιδέα να ζητήσουμε ελέγχου, ε, κάτι το οποίο εκπλήρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν πάρα πολύ επιτυχη η προσπάθεια προσπάθεια γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας για περισσότερους ελέγχους στο, στην αεροπο, για την αερο, αεροδρόμια ε, και έτσι βοήθησε πάρα πολύ τις εθνικές αρχές. Ξέρετε ότι... Είναι κάτι το οποίο, στο οποίο όλες οι χώρες ε, συμφώνησαν οι περισσότερες τουλάχιστον, εκτός από την πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνετε εσείς να μας διατηρείτε ασφαλείς, ε, έχουμε και τον εμπειρογνώμονα από, το, από τη CIA, ε, φαντάζομαι θα γνωρίζεστε, ε, η αντι κατασκοπία είναι κάτι το οποίο έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των ταξιδιωτών, οπότε πιστεύω ότι πρέπει ε, όλων τις προσπάθειες να τις επενέσουμε και των μεν και των δε. Έχει πάει πάρα πολύ καλά η προσπάθεια. Υπάρχουν όμως κάποια ζητήματα. Αναφερθήκατε στα υγρά. Πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για τις συζητήσεις περασμένης εβδομάδας, εμένα Εμένα, εγώ πάντοτε έλεγα, ας είναι η τεχνολογία σωστή ώστε να δουλεύει, αλλά εντάξει, τουλάχιστον ας κρατήσουμε τα 100 ml, γιατί Δυστυχώ με αυτό πρέπει να μείνουμε. Πάντως οι Αμερικάνοι πιστεύουν ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Αν χρειάζεται λοιπόν για τη διαμετακόμιση θα χρειαστούν επιπλέον έλεγχοι ή αλλαγές. Δεν νομίζω όμως ότι καταλαβαίνει κανείς ε, τι σημαίνει όλη αυτή η αλλαγε δεν νομιζω ομως οτι καταλαβαινει κανεις τι σημαινει ολη αυτη η διαδικασια των 100 ml και αν κάνουμε λίγο περισσότερε συζητήσει, θα γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Ήταν πάρα πολύ πρόημο να καταλήξουμε σε μία ε, ε, απόφαση για τα υγρά. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και πριν από χρόνια όταν καταλήξαμε στα 100 ml. Εγώ δεν είμαι απεσιόδοξη. Αυτό ήταν ε, αυτό ήταν ο στόχο τη προσπάθεια, ότι μπορεί σε γενικές γραμμές ε, να δουλεύει σε κάποιες χώρε. Ε, αν δεν είναι κανεί στη Σέγγεν, ούτως ή άλλως περνάει από πάρα πολλού ελέγχου ασφαλεία. Ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί αυτή η αλλω περναει απο παρα πολλού ελέγχου ασφαλεία. ελπιζουμε οτι θα βελτιωθει αυτη η κατασταση σε γενικές γραμμές λοιπόν νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει. Απλώς θα ήθελα ε, ως τελευταίο σημείο να πω το εξής. Επειδή εγώ δούλευα σε αεροπορικέ εταιρείε και πραγματικά παίρνω πολύ σοβαρά το θέμα τη ασφάλεια, πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπω έχουν τα πράγματα τώρα. Ε, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Πάρα πολύ καλό είναι ότι οι επιστήμονες λένε υπάρχει πολύ καινούργια τεχνολογία κλπ. Είναι πολύ άσχημη η εμπειρία των επιβατών και δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Οι τρομοκράτες ε, γίνονται και αυτοί πολύ πιο εξελιγμένοι, εξελίσσονται. Πρέπει να σκεφτούμε και διαφορετικά. Το θέμα είναι να βασιζόμαστε στον κίνδυνο. 99,999% όλοι αυτοί οι άνθρωποι και εμείς εδώ μέσα δεν έχουμε κανένα σκοπό να βλάψουμε κανέναν. Δεν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Πρέπει να πω ότι όλο αυτό το σύστημα των ε, εκ των προτέρων ελέγχων που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή ε, ε, στις ΗΠΑ μας δείχνει πώς πρέπει να κινηθούμε. Δεν λέω να γίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί είναι κάτι το πολύ μαζικό. Πρέπει να γίνει αναχώρα. Αλλά αν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι επιμένουν πάρα πολύ στην ασφάλεια, όπως γνωρίζετε, θεωρούν ότι αυτός είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε και ο κόσμος θέλει να το αποδεχθεί αυτό. Αν εγώ θέλω να σα δώσω περισσότερες πληροφορίες, ε, αλλά περνάω λίγο πιο γρήγορα από τον έλεγχο, τόσο το καλύτερο για μένα να σας πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι για τακτικούς επιβάτες πρέπει να βρούμε διαφορετικό τρόπο ελέγχου, γιατί αλλιώς θα πρέπει να περνάμε από body scan για να πάμε στο Manchester από εδώ. Και το βρίσκω πολύ προβληματικό αυτό και δεν θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πείτε μας ε, και σε εμά και στους υπουργούς εσωτερικών μας, σε όλους, ότι βλέπουμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά για το πώς θα αξιολογούμε τον κίνδυνο. Ε, έχουμε τον Ήρα ως απειλή σε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ε, δεν σημαίνει ότι κάθε Ιρλανδός είναι τρομοκράτης. Καταφέραμε όμως να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να σκεφτούμε διαφορετικά για το ISIS. Πρέπει να σκεφτούμε απλά διαφορετικά γενικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την ενημέρωση. Προφανώς θα γίνει αναθεώρηση. Μιλήσαμε με τον Επίτροπο. Ε, συμφωνούν, ε, συμμετέχουν γιατί νομίζω ότι θέλουν να έχουν μεγαλύτερο ρόλο και αυτό είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους της ομάδας μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Έχω πολλές παρατηρήσεις όμως, πολλές ερωτήσεις. Πού μπορούμε να εξασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων, των ιδιωτικών, όταν ε, υπάρχουν προσωπικά στοιχεία που δίδονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου και το ίδιο γίνεται και με τους επιβάτες και με, τους, και με τα αεροπλάνα που μεταφέρουν εμπορεύματα. Αυτές οι νέες ε, προσεγγίσεις των μέτρων ασφαλείας ε, και όλα αυτά τα μέτρα που προκύπτουν γίνονται σε πλαίσιο εγγύησης αποτελεσματικότητας και τι γίνεται με τις αποσκευές ε, που μπαίνουν στο αεροσκάφος, που σκανάρονται και ελέγχονται. Ποιο είναι το κόστος και το κόστος αυτό το, το επιβαρύνει μόνο τα αεροδρόμια. Και δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί το όλο σύστημα αν κάποιος ε, περνάει τις αποσκευέ του από τσεκίν. Ο κύριος Γιούνκερ για παράδειγμα έχει ένα κουτί σοκολατάκια και μία κονσέρβα μέσα στην αποσκευή του. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν ή ο κύριος Γιούνκερ έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ότι αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται κάποιοι και για ποιο χρονικό διάστημα. Αυτές είναι πραγματικές ε, ερωτήσεις, ε, πραγματικά ζητήματα σήμερα και ε, αυτά είναι που πρέπει να μας οδηγήσουν στο να καταλάβουμε πώς πρέπει να δράσουμε. Ο Γιάννης έχει το λόγο. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση. Ήταν πολύ καλή. Θα ήταν καλό να την έχω και σε ηλεκτρονική μορφή για να την κρατήσω. Μπορώ να το ρυθμίσουμε ίσως. Είναι αρκετά δύσκολο να δω ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προς ποιος της υπηρεσίας. Έχω μία ερώτηση που θα αναφέρω αργότερα. Θέλω να αναφερθώ στη στρατηγική και τη συμπερίληψη των πτυχών ασφαλείας και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που έχω αναφέρει και εδώ στις εσωτερικές πτήσεις που υπόκειται σε, προμήθ... διαγωνισμούς στη Σουηδία. Σημαντικές διαδρομές που πηγαίνουν σε πόλεις με μεγάλα νοσοκομεία, πολύ σημαντικό θέμα όταν γίνεται διαγωνισμός για αυτές τις διαδρομές και έχουμε στονική εταιρεία που αναλαμβάνει αυτό το δρομολόγιο και μετά οι Σουηδικές αρχές είναι υπεύθυνε για την ασφάλεια. Και μετά από διάφορα γεγονότα διαπιστώνουν ότι η αεροπορική εταιρεία θα έπρεπε να απαγορευτεί, να μην επιτραπεί να πετάξει. Αλλά οι Σουηδικές αρχές δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Οι Ιστονικές αρχές θα πρέπει να απαγορεύσουν τις πτήσεις, διότι εκεί έχει την έδρα της η εταιρεία. Αλλά δεν το γνωρίζουν και αν το γνωρίζουν δεν λένε κάτι γιατί λένε δεν θα αποφασίσουμε επί απαγορεύσεως. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός δεν κάνει τίποτα. Άρα τελικά δεν γίνεται αλλαγή. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το σύστημα. Ό, όταν γίνονται οι έλεγχοι και διαπιστωθεί ότι πρέπει να απαγορευτεί αεροσκάφος ή εταιρεία, ε, διότι υπάρχουν προβλήματα με την ασφάλεια κλπ. Και, και υπάρχει άλλη αρχή σε άλλη χώρα που λέει δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τι πτήσει. Υπάρχει συστημικό πρόβλημα εδώ. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε αυτό. Για την ώρα έχουμε μια εταιρεία η οποία λειτουργεί για εσωτερικέ πτήσει στη Σουηδία, την μποϊκοτάρει ο κόσμος, προτιμούν να πάρουν λεωφορείο και να κάνουν 400-500 χιλιόμετρα και μποϊκοτάρουν και επιχειρήσουν την εταιρεία, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Επιτέλους έχει το λόγο ο George Bach. Ευχαριστώ. Μην έχετε μεγάλες προσδοκίες όμως από αυτά που θα πω. Όχι, αστείευομαι. Χαίρομαι και ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίαση. Δύο-τρία ερωτήματα θέλω να θέσω. Όσον αφορά την ευελιξία, είπατε και δικαίως ότι στους ε, ελέγχους ασφαλείας τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που αποφασίζουν τις μεθόδους. Ξέρω όμως από προσωπική εμπειρία ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί τελικά ανασφάλεια στους επιβάτες ε, Υπάρχουν διάφορα μέτρα που εφαρμόζονται σε διάφορα αεροδρόμια, κάτι που επιτρεπόταν πέρσι δεν επιτρέπεται πια και νομίζω ότι από αυτή την άποψη αυτή η ευελιξία μάλλον δεν είναι και τόσο πλέον Πείτε μας, εσείς γιατί θεωρείτε ότι είναι πλέον η ε, ευελιξία αυτή. Επίσης, όλα αυτά αφορούν και το προσωπικό. Το προσωπικό εδάφους, το προσωπικό αέρος, τους πιλότους, την μετεκπαίδευσή τους, την κατάρτισή τους. Και, αυτό, και όλα αυτά τα θέματα εμπίπτουν ε, ε εντός αυτής της ευελιξίας. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν δηλαδή τι θα κάνουν. Και τελευταίο, ε, ως ευρωβουλευτές πολλές φορές παρακολουθούμε και ενημερωνόμαστε από την πλευρά του κλάδου ε, και υπάρχουν ε, διάφορες προτάσεις. Πόσο σοβαρές είναι αυτές, πώς μπορούν να καταστούν πιο αποδοτικές αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις ε, με τους σαρωτές, μήπως τελικά αν υπάρξουν επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες ε, διαπιστώσουμε μετά από 6 ή 12 μήνες ότι ε, τελικά δεν ήταν και πολύ σωστή η επένδυση αυτή επειδή ξεπεράστηκε από τις ίδιες τεχνολογικές εξελίξεις. Ποια, ποια, ποια είναι η άποψή σας για την συνεργασία με τον κλάδο. Πρόεδρος, και εγώ έχω ένα ερώτημα για τα υγρά. Είχαμε κάνει συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή και μάλιστα και, και κλεισμένων ε, των θυρών και δεν μας απάντησε κανείς ποια τελικά, ποιος είναι τελικά ο λόγος. Εμείς ζητήσαμε την, ε, ζητήσαμε την κατάργηση αυτής, την άρση αυτής της απαγόρευσης. Θεωρήσαμε δε ότι υπάρχει, είναι, ένας, είναι ένας κρυμμένος τρόπος ε, επιχορήγησης των ε, duty free είναι πάρα πολύ απλό. Αφού τελικά επιτρέπεται, 100, ε, επιτρέπονται 100 ml, μπορούν 3-4 ε, ε, τρομοκράτες να χωρίσουν την αναγκαία ποσότητα και να βρεθούν στο αεροσκάφο και τελικά να κάνουν. Ή, για παράδειγμα, να πάρω, ε, χρειάζομαι ένα εκρηκτικό υγρό που αποτελείται από ένα υγρό και μια σκόνη και ο ένας παίρνει τη σκόνη και ο άλλος παίρνει το, το, το υγρό και, και δημιουργώ τελικά ε, το εκρηκτικό αυτό υγρό πάνω στο αεροσκάφος. Μπορείτε να μας πείτε τελικά ποιος ήταν ο λόγος που έγιναν όλα αυτά. Έγινε κάτι γιατί έπρεπε να απαντήσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο κίνδυνο. Έχετε κάποια ανάλυση. Ποια είναι αυτή. Γιατί εδώ και χρόνια ακούμε ε, ότι θα υπάρξουν τεχνολογικές εξελίξεις με τις οποίες θα μπορέσουμε να ε, εντοπίζουμε την επικινδυνότητα συγκεκριμένων υγρών. Αλλά πείτε μας, σας παρακαλώ, επιτέλους, ε, ποια είναι η ανάλυση σας ή παραδεχτείτε ότι επρόκειτο για λάθος και ότι ε, θα άρουμε τη συγκεκριμένη απαγόρευση και θα, θα λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Έχετε το λόγο κύριε ο Και οι Αμερικάνοι πάντως μου είπαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ε, ε απολύτως εφικτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση. Πράγματι δεν έχουμε 60.000 άτομα όπως η TSA και το Ευρωπαϊκό Σύστημα βασίζεται κατά πολύ στην αλυσίδα της επικουρικότητας βασιζόμαστε κατά πολύ στα κράτη-μέλη και τις αρχές των κρατών μελών. Παίζουμε το ρόλο του παρόχου των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη με μια εξαίρεση αξιοσημείωτη με το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά ποια ήταν η βασική ιδέα να διαφυλάξουμε το βασικό δηλαδή την εσωτερική αγορά. Μπορείτε να φανταστείτε στο σημερινό κόσμο της αεροπορίας με τις διαλέψεις που έχουμε αν δεν είχαμε ένα σύστημα εμίας μίας εξέτασης ε, χειραποσκευών που θα αναγνωρίζεται από κάθε χώρα. Θα γινόταν ε, η έλεγχη σε κάθε σημείο. Θα ήταν χάος τα αεροδρόμια και πολύ δαπανηρό και για αυτό. Γι' αυτό το όλο σύστημα βασίζεται όχι μόνο επί των αρχών των κρατών μελών που διαθέτουν τα περισσότερα μέσα για την ασφάλεια, αλλά βασίζεται και στη συλλογή πληροφοριών. Δεν έχουμε φτάσει, και σωστά το είπε κυρία Φώστερ, ότι χάρη στις εθνικές αρχές μπορούμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες και μπορούμε να τι αναλύσουμε. Τα τελευταία χρόνια το σύστημα βελτιώθηκε δραματικά. Και η προθυμία όλων των κρατών μελών να μοιράζονται τι πληροφορίε παίζει ρόλο για τη βελτίωση του συστήματος. Είναι θετικότατη εξέλιξη. Βάσει των πληροφοριών αυτών καθορίζουμε από κοινού με τις εθνικές αρχές τα βέλτιστα προς εφαρμογή μέτρα. Και με μια άλλη ιδέα που μαχητικά υπερασπίστηκε η κυρία Φώστερ. Να έχουμε έναν μικρό πυρήνα επιθεωρητών που εξασφαλίζουν την εφαρμογή των μέτρων. Παντού. Με το ίδιο ποιοτικό επίπεδο σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε πλήρη συνεργασία το κάνουμε αυτό με τις εθνικές αρχές. Δεν χρειάστηκε να δημιουργήσουμε στρατιά επιθεωρητών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως για θέματα πυρηνικής ασφαλείας. Βασιζόμαστε στους πόρους των εθνικών αρχών των κατών μελών. Τέλος. Όσον αφορά τα διάφορα μέτρα που αναφέρατε σε σχέση με τη διευκόλυνση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επιβατών. Υπάρχουν ιδέες που θέλουμε να αναπτύξουμε στην επερχόμενη στρατηγική για τις αερομεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα σας υποβληθεί. Θέλουμε να προχωρήσουμε όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση με διάφορες χώρες δεν έχουμε πετύχει το πλήρες δυναμικό που θα μπορούσαμε και οι συζητήσεις με τις ίπα πάνω σε αυτό το έδειχναν. Υπάρχει κάποια αντίσταση ακόμα, αλλά πολύ καλύτερη κατανόηση όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος και όσον αφορά το επίπεδο που έχουμε πετύχει, όπως είπε ο Κάλλος, πόρο απέχουμε από τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΙΚΑΟ και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Δεύτερον, η εκ των προτέρων έγκριση, το θέμα αυτό που αναφέρατε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε σοβαρά, διότι εάν υπάρχει αυτή η πρώτερη έγκριση σημαίνει ότι είμαστε σοβαροί για την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων ασφαλείας και μέσω της πρόθεσης της πρώτερης έγκρισης από τις ΙΠΑ θα βελτιώσουμε δραματικά το βαθμό της αμοιβαία αναγνώρισης. Και πράγματι, αν εφαρμοστεί σωστά στα αεροδρόμια, θα είναι η καλύτερη ποιοτική βελτίωση για το ταξίδι των επιβατών. Και αυτό θα είναι κάτι που έχει πολλά χρόνια να γίνει. Και αυτό θα ήθελε να προωθήσει η Ευρώπη και να προωθηθεί και σε άλλες χώρες βάσει της ε, επιτευχής σας εμπειρίας. Μετά, τεχνολογία, πολύ το θέσατε, η τεχνολογία πράγματι υπάρχει για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων και ελπίζουμε βέβαια και για τη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών. Πρώτα απ' όλα για τα υγρά, κύριε Πρόεδρε, σήμερα μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν ήταν ανόητη ιδέα να κινηθούμε όσον αφορά τα υγρά. Καθόλου. Και αν έχουμε ακόμα την απαγόρευση για τα υγρά, έχουμε στοιχεία. Συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία. Μπορώ να σας πω ότι ίσως κάναμε ένα λάθος να υποσχεστούμε κάποια προθεσμία. Δεν ήταν καλή ιδέα αυτή πιθανότατα. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, να δούμε το τι μπορεί να πετύχει τεχνολογία, το είδος της απειλής και μετά εν ευθέτω χρόνο να κάνουμε πρόταση. Αυτό που κάνουμε για τα υγρά είναι πρωτίστως να επιβεβαιώσουμε νέου ότι ο στόχος μας όπως είπε και ο Κάρλος είναι να παραμείνει η απαγόρευση Μάλλον να αρθεί απαγόρευση, αλλά πρέπει να πληρούνται οι προποθέσει. Πρώτη προπόθεση, να υπάρχει τεχνολογία, η σωστή που θα χρησιμοποιείται σε όλα τα αεροδρόμια. Και η τεχνολογία να μα το επιτρέψει. Όπω είπε η κυρία Φώστερ, Πιθανότατα πρώτο βήμα θα ήταν όταν θα υφίσταται η τεχνολογία να βρούμε ένα σύστημα που θα βασίζεται στην επιλογή των επιβατών. Πολύ σημαντικό και σταδιακά να το χρησιμοποιήσουμε για όλους επιβάτες. Είμαστε πολύ σοβαροί γι' αυτό όμως. Και τακτικά και οι τρεις άλλες σημαντικές χώρες στον κόσμο έχουν δεσμευτεί να μας βοηθήσουν. Η ΙΠΑ, η Αυστραλία και ο Καναδάς. Και να παραμείνουν στις υποσχέσεις τους. Παρά κάποιο σκεπτικισμό που επικρατεί καμιά φορά. Το έχετε συζητήσει αυτό στη ΣΥΠΑ. Ο ρόλος της ΕΑΖΑ, άπρος ενδιαφέρον θέμα. Ξεκινήσαμε μια μελέτη. Θα μας βοηθήσει αυτή να συναγάγουμε ενδεχομένως συμπεράσματα περί ενδεχομένων βελτιώσεων στον τομέα της ασφαλείας, στα πλαίσια της ΕΑΣΑ, αλλά υπάρχει και περιθώριο για εργασίες και προσπάθειες εκεί. Ίσως μπορέσουμε να βελτιώσουμε το γενικό σύστημα που διαθέτουμε. Τέλος, όσον αφορά τον έλεγχο των αποσκευών, ο έλεγχος αποσκευών για χειραποσκευές και όλα ε, γενικά τις επισκευές είναι διαφορετικές. Καμία πληροφορία δεν κρατείται απαντώ στην προκλητική ερώτηση ενός βουλευτού όσον αφορά το μπουκάλι του κονιάκ. Δεν θα υπάρχει τέτοιο αρχείο που θα ταυτίζει έναν επιβάτη με τα όσα βρίσκονται στη βαλίτσα του, βαλίτσα τη ανεξάρτητα από το τι είδους ε, αποσκευή είναι, αλλά λειτουργεί καλά το σύστημα του ελέγχου των αποσκευών, χρησιμοποιείται άριστη τεχνολογία σε όλα τα αεροδρόμια, 100% έλεγχος γίνεται ο, ε, όσον αφορά τι αποσκευέ, χειραποσκευέ, αποσκευέ καμπίνα, ε, βελτιώνεται η κατάσταση. Θα δείτε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο ότι πράγματι τα αεροδρόμια όλο και περισσότερο θα χρησιμοποιούν την ανείχνευση εκρηκτικών για να ελέγχουν και τις χειραποσκευές και τις αποσκευές καμπίνας και θα μπορούν να προβούν στην αναγκαία ανάλυση για νέες απειλές. Η άλλη ερώτηση που αφορά την εστονική αεροπορική εταιρεία που δεν γνώριζα. Αυτό σχετίζεται με την ασφάλεια που θέσατε. Όσον αφορά την ασφάλεια υπάρχουν μηχανισμοί να μπορούμε να δράσουμε όταν μια εταιρεία δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ασφαλείας. Όχι μόνο η ΕΑΖΑ, ο φορέας, αλλά υπάρχει και ευρωπαϊκός μηχανισμός που μπορεί να κινηθεί. Θα το παραπέμψω στους συναδέλφους υπευθύνου για την ασφάλεια και θα έρθω σε επαφή και με τις εστονικές και σουηδικές αρχές να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, διότι κανονικά υπάρχει άμεση ροή ε, πληροφοριών και αν δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας μιας εταιρεία, τις απαγορεύονται πτήσεις αμέσως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Νίδη. Μια τελευταία σημείωση. Στις 12.30 θα ξεκινήσει εδώ στην αίθουσα ένα σεμινάριο ε, από την ε, Γενική Διεύθυνση MOVE για το πακέτο Juncker. Είναι, είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να παραμείνετε εδώ, να δείτε, να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς, ιδιαίτερα τους συναδέλφους από την ε, πορτογαλική καμπίνα που τους γνωρίζω και προσωπικά. Γεια σας και θα τα πούμε στις τρεις